Uh, Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Αν έχετε την καλοσύνη. And, I... <laughs> Και όπως είπε σχέθηνε χθες, αρχίζουμε τις ψηφοφορίες μας επακριβώς στις 9 το πρωί. Αλλά έχασα, έχασα το στίχημα τον εαυτό μου. Ένα λεπτό μετά τις 9 είναι και ξεκινάμε. Την άλλη φορά μου θα είμαι ακόμα πιο αυστηρό, σας το υπόσχομαι. Ε, βάση περιπτώσει, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσουμε. Την ψηφοφορία θα ξεκινήσουμε την έκθεση Bauer. εφαρμογή τη ισότητα τη αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία τη αυτή αξία. Ξεκινούμε λοιπόν. Είσαστε έτοιμοι όλοι και όλε. Λίγο πιο ήρεμα παρακαλώ μόνο. Αν μπορούμε. Κυρία Γιανακουλάκη. Please be a little bit calmer inside here when we vote. Λίγη ησυχία παρακαλώ για να ξεκινήσουμε. Τροπολογία. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Λάθος ε, πρώτη της απασχόλησης υπέρ. Κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Πρώτη της απασχόλησης. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Okay, we have to check that once again. Να το ξαναδούμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απέριφθη. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το επαληθεύσουμε. 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται προφανώς. 35 καταπίπτει. Όχι. Λυπούμε, διορθώνω. 35 την ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 15 της απασχόλησης. Κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ. Κατά αποχές Ας το επαληθεύσω όμως 37. Ναι, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε ψηφοφορία. Απερίφθη. 36 κατά αποχές εγκρίνεται. 38 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Απορρίπτεται νομίζω. Ας επαληθεύσουμε όμως τη 40, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 41 περίφθη. Πάμε στην... Ε, έχει απορριωσευθεί μάλλον 43 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 44 υπέρ, κατά ε, αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται μάλλον. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 46 και 47 της απασχόλησης καταπίπτουν. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 47 και 40 της απασχόλησης καταπίπτουν. 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. 51 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ήταν μάλλον αμφιλεγόμενο το αποτέλεσμα. Στο δεύτερο τμήμα λοιπόν της 51 άρχισε η ψηφοφορία, η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 καταπίπτει. Συμβαστική 12 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 53 καταπίπτει, η 35 της απασχόλησης δεν θα ψηφίσει στο πρώτο και το δεύτερο τμήμα. Και να πάμε στη 48, υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται, 36 καταπίπτει, 54, 54 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, έκτη της απασχόλησης υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 19 της απασχόλησης υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13-14 δεν 16 υπέρ της απασχόλησης κατά αποχές ας το επαληθεύσουμε 16 της Επιτροπής Απασχόλησης παρακαλώ Άρχιτη ψηφοφορία πέρασε Απορρίπτεται. 28, οι 34, 33 της Επιτροπής Απασχόλησης δεν θα ψηφιστούν. Η ε, ε, τροπολογία 50 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Ας επαληθεύσουμε την 50 της Επιτροπής Απασχόλησης. 50 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και μετά έχουμε μια σειρά από τροπολογίες Επιτροπής Απασχόλησης που δεν θα ψηφιστούν. Και προχωρώ στην 53 της Επιτροπής Απασχόλησης. 53 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και στη συνέχεια πολλές της Επιτροπής επασχόλησης που θα ψηφιστούν και πάμε στην 56 υπέρ κατά αποχές το νομίζω 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 58 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 59 υπέρ να επαληθεύσουμε την 58 καλώς 58 επαλήθευση άρχη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται <laughs> Έχω και καινούρια γυαλιά σήμερα, να ξέρετε. Πέρας της προφορίας. Άρα εγκρίνεται ε, η 13 συμβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 60 καταπίπτει, 14 υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται, η 61 καταπίπτει, 62 υπέρ, κατά αποχές. Όχι, δύσκολο, δύσκολο να το παρακολουθήσουμε. Επαληθεύουμε την 62 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 Προφορική τροπολογία. 65 υπέρ λοιπόν. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ, υπέρ της 67 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται, 68 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται, 37 δεν ψηφίζεται, δεν υπέρ απασχόληση. 69 υπέρ, κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε την 69 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 21 και 25 της απασχόλησης δεν ψηφίζονται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 73 καταπίπτει 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 έχει αποσυρθεί 79 τώρα υπέρ κατά αποχές Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές Πάμε τώρα, η 80 καταπίπτει, πάμε στην 5 της απασχόλησης που θα ψηφιστεί, 52 υπέρ, κατά αποχές, νομίζω ότι πρέπει να επαληθεύσουμε. 52α της απασχόλησης, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Και έτσι ψηφίζουμε την υπαριθμόν 81 υπέρ, κατά, αποχές. Απερίφθη. 82 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 4, 24, 26 και 27 της Επιτροπής Απασχόλησης δεν ψηφίζονται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 83 υπέρ, κατά αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη. Ας παληθεύσουμε την 83 άρχιτη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 C και 52D της απασχόλησης δεν ψηφίζονται. Ψηφίζουμε την 52B υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 52F σιγματάφ της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και προχωρούμε έως την 85, 85 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 18 της απασχόλησης ψηφίζεται, η 86, παρακαλώ τώρα, τροπολογία 86, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται να επαληθεύσουμε το 87. Εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές. Δεν μπορούσα να διακρίνω το αποτέλεσμα. Παρακαλώ να επαληθεύσουμε την 88 υπέρ. Μάλλον άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. 89 και 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 11 και 20 της απασχόλησης τα ψηφίζονται. 23 της Επιτροπής Απασχόλησης παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμόν 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3, 4, 5 καταπίπτουν. Συμβαστική υπαριθμόν 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 6 και 7 καταπίπτει. Και πάμε στην 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 της απασχόλησης θα ψηφιστεί. 9 ε, ναι, παρακαλώ υπέρ, κατά αποχές Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε τη 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Απερίφθη. 13 υπέρ κατά άποχες απερίφθη 14 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε τη 14 άρχεται η ψηφοφορία τροπολογία 14 Πέρα τη ψηφοφορία. Just closed. It's rejecting clearly, but it, you did... Πέρασε ψηφοφορίας, αλλά δεν είχατε σηκώσει και το χέρι, έτσι, ε, απερίφθη. Συμβαστική τρία. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Δεκαεννέα. Δεκαπέντε. 30 και 29 της απασχόλησης καταπίπτουν και πάμε στην συμβαστική παριθμών 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 16 8 9, 10 της απασχόλησης και 17 καταπίπτουν. Πάμε στην 3 της απασχόλησης. Μόνο όμως... Α, όχι, και αυτό καλύπτεται. Επομένως πάμε στη 18, τροπολογία υπερθυμών 18, υπέρ. Κατά αποχές. Δύσκολο να διακρίνω αποτέλεσμα. Ας επαληθεύσουμε τη 18. Απερίφθη νομίζω, αλλά ας επαληθεύσουμε. Πέρα στις ψηφορίες. Απερίφθη. Τροπολογία 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 άλλες δεν έχουν αποσυρθεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ψηφίσουμε τότε την 25 σας παρακαλώ σας παρακαλώ αν έχετε κάτι να συζητήσετε παρακαλώ έξω την αίθουσα Ψηφίζουμε την 25 τώρα, παρακαλώ, τροπολογία 25, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε την 25, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. Ε, συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 26 καταπίπτει και η 31 της απασχόλησης επίσης. Πάμε στην 27 υπέρ κατά αποχές Να επαληθεύσουμε την 27. Άρχεται η ψηφοφορία για την 27. The vote Has Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 29 υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να επαληθεύσουμε την 29, αρχή ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13, 31 ε, κατά 30-31 μάλλον καταπίπτουν. Περ κατά αποχές εγκρίνεται 2 περ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε τώρα στο σύνολο του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Λείπει μία ψήφος μάλλον. Πέρα στις ψηφοφορίες. 28 εγκρίνεται προφανώς και συγχαρητήρια.

Να περάσουμε στο επόμενο σημείο στον κατάλογο των ψηφοφοριών. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί ε, το κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων και το καθεστώ που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζουμε την ψηφοφορία με τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά η κρίνεται. 21 υπέρ. Με συγχωρείτε. Δεν είναι στον καταλογό μου. Λοιπόν, τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε την 3. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 3. Has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Σε δύο τμήματα. Χωριστή ψηφοφορία. Τηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να ελέγξουμε την 6 νομίζω, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 6. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Και αυτό σημαίνει ότι καταπεπτεί 8 και παίρνουμε στην 9 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 26 καταπίπτει, παίρνουμε στην 27 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 25 καταπίπτει. Τροπολογία 29 ναι, υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 30 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά Αρχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. είδατε, η 12. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 35 και 36 καταπίπτουν. Περνάμε στην 37 και στην 38. Είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά, εποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 14, υπέρ, κατά, εποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 15, υπέρ, κατά, εποχέ. απορρίπτεται. Τροπολογία 16, υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 17, υπέρ, κατά, μπουχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. μπουχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. μπουχές Απορρίπτεται. Και θα ψηφίσουμε ένα μέρος της τροπολογίας 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου, άρχεται η ψηφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Με 20 υπέρ. 5 ψήφους κατά. Χαρητήρια για την εισηγητρή. We then, uh, we then vote on the next. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Αλία μικρή κλίμακα και παραδοσιακή ελεία και μεταρρύθμιση της κοινωνικής πολιτική. during the voting, I really want you to, to be very silent because. Θα ήθελα να υπάρχει ησυχία κατά τη διάρκεια της ψηφοφορία. διαφορετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για του βουλευτέ να ακούσουν τι λένε. Και εγώ είμαι εδώ για σας. Τροπολογία 12. Θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία με την τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 και 14, οι τροπολογίες αυτές καταπίπτουν. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, εποχέ. εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, εποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά εποχές πρέπει να ελέγξουμε νομίζω την τροπολογία 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Απολογία 24 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 και 26 καταπίπτουν, τροπολογία 29 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 3 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 18-19 καταπίπτουν, το συμβιβασμό 4 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22, 32 και 33 καταπίπτουν, συμβαστική οι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα περάσουμε στην 34 υπέρ κατά αποχές πολύ δύσκολο να δούμε το αποτέλεσμα να ελέγξουμε την 34 άρχεται η ψηφορία την 34 μέρες Εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι τροπολογίε 2 και 4 καταπίπτουν και πάμε στην τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αγωχές, νομίζω εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αγωχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αγωχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. εποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. εποχές, Εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε το σημείο του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. vote is closed. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια. Uh, next, oh, sorry. Uh, next, next item is. Επόμενο σημείο. Ερώτηση για κανονισμό του Συμβουλίου για το εφαρμοστό δίκαιο στι αποφάσει σχετικά με τι περιουσιακέ σχέσει μεταξύ των συζύγων. Ξεκινάμε την τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 31, υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε την 7, υπέρ, κατά, αποχέ, να ελέγξουμε την 7, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι είναι δύσκολο να δούμε το αποτέλεσμα. Να ελέγξουμε λοιπόν την τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Λοιπόν, πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας, γιατί φορτικά θα πρέπει να ψηφίζουμε για κάθε σημείο, γιατί δεν είμαι σίγουρος και καθυστερούμε. Σας παρακαλώ, λοιπόν. Και κυρία Ταμψόν, δεν θα τα κάνω έτσι γρήγορα, γιατί θέλω όλοι να ξέρουν τι συμβαίνει, ακόμη και αν σας γνωρίζετε τι συμβαίνει. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν για τροπολογία 8. Πέρας. Εγκρίνεται. Βλέπετε, αν δεν μπορώ εγώ να διακρίνω, εσείς πρέπει να σηκώσετε το χέρι. Λοιπόν, τροπολογία 32. Υπέρ, κατά, εποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Νομίζω. Και αυτό σημαίνει θα το ψηφίσω μόνο ένα τμήμα. Η τροπολογία 35, ένα τμήμα λοιπόν της 35 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 35, το τμήμα της 35, άρχεται η ψηφοφορία. 35. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές υπέρ 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε και 12. Να ελέγξουμε τροπολογία 12. No? Okay. Then we count. I uh, will check on amendment 2. Να ελέγξουμε τη 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. It's rejected. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Επιτυχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Λέω να ελέγξουμε τα 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μα είναι αδύνατον. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Εποχές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 εποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη. 26 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, ελέγξουμε την 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεν θα ψηφίσουμε την 1. Υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Με συγχωρείτε ψήφισαμε την 1. 29. Υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, εποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, εποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Να αλλάξουμε την 30. Την τροπολογία περιθμών 30, έρχεται ψηφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ. Κατά. Εποχές, εγκρίνεται και να ψήσουμε στο... για το σύνολο της γνωμοδότησης, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην συγγήτρια. Next findings is the proposal. Επόμενη πρόταση για την υγεία και την ανάπτυξη, τρίτο πολιετέ πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020 και να σας ρωτήσω, θα μπορούσαμε να τα ψηφίσουμε όλα μαζί, unblock. Όχι την πρώτη μόνο, όχι. Εντάξει. Ωραία, να ψηφίσουμε λοιπόν την πρώτη και μετά τι υπόλοιπε. Πρώτη τροπολογία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και Τώρα να ψηφίσουμε όλες τις υπόλοιπες μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εγκρίνονται μάλλον. Πρόταση για τον κανονισμό λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέσω του Να ψηφίσουμε όλοι μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέσου σταθερότητα, παρακαλώ. Να τα ψηφίσουμε όλα μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση έχει στην κρίση. Και αυτά θα τα ψηφίσουμε μαζί. Το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Να ψηφίσουμε λοιπόν όλα εκτός από την τροπολογία 1 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή.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

θα το γυρίσω στο Σουηδικά, αλλά να ξέρετε ότι θα επιστρέψουμε σε ένα ε, θέμα το οποίο αναβάλαμε για σήμερα από χτες για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας. Αν θέλετε λοιπόν να ηρεμήσετε λίγο, στις 10.30 θα έρθει εδώ η Επίτροπος Ρέντινγκ. Έχουμε 40 λεπτά. Αλλά πρώτα θα συζητήσουμε το 7 της ε, ημερήσιας διάταξης. Το λόγο έχει η κυρία Μποσκούρτ. Και σας παρακαλώ λίγο πιο ήσυχα. Αν θέλετε να μιλήσετε, βγείτε έξω. Ευχαριστώ. Thank you, dear Chair. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε για το θέμα αυτό, για την ε, νέα πρόταση που μας ε, υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς αλλάζουν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, τους, ε, με τις γειτονικέ χώρες. Η νέα αυτή η προσέγγιση θα υποστηρίξει τις, τα κοινοβούλια που υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις και τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη απόδοση ευθυνών. Και στο μέλλον το ευρωπαϊκό αυτό μέσο ε, μηχανισμού γειτονίας θα συνδέεται με το ευρωπαϊκό όραμα Είμαι σε διαρκή επαφή με τις γυναίκες της Αραβικής Άναξης και μας δηλώνουν ότι χρειάζονται βοήθεια σε ό,τι αφορά την διοργάνωση των προσπαθειών τους και ότι χρειάζονται βοήθεια από τους ομολόγους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν έδωσα ιδιαίτερη προσοχή για την οικοδόμηση ε, σχέσεων μεταξύ των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Αραβικής Άνοιξης. Δέκα τροπολογίες έχουμε συνολικά. Οι δικές μου τροπολογίες καταστούν σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών προκειμένου να τονωθούν οι γυναίκες ε, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους και στην αγορά εργασία και στις πολιτικές θέσεις λήψης αποφάσεων, μηδενική ανοχή ε, σε ό,τι αφορά τη βία κατά των γυναικών, προστασία των γυναικών που είναι θύματα βίας, αντιμετώπιση θεμάτων ατιμορρησίας, ε, καταπολέμηση του τράφικινγκ, καταπολέμηση των ε, εξαναγκασμένων γάμων, λοιπόν, προώθηση της ε, κοινωνίας των πολιτών και των γυναικείων οργανώσεων και γενικά mainstreaming σε θέματα που αφορούν τα δύο φύλλα. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω και αναμένω τις παρατηρήσεις σας. Thank you very much for that. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα μιλήσω σου ειδικά τώρα πια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Αν έχετε σχόλια, παρατηρήσεις, τώρα είναι η στιγμή. Δεν φαίνεται να υπάρχουν παρατηρήσεις λοιπόν, δεν ζητά κανείς το λόγο. Okay. Θέλει κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως να πάρει το λόγο. ovanligt. I, i sådana fall så får jag helt enkelt bara... Μάλιστα. Να ρωτήσω μήπως θέλει η κυρία Ποσκούρτ να συμβουλεύσει κάτι. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, να πω μόνο ότι ελπίζω ότι αυτό αποτελεί μια ένδειξη ότι όλοι υποστηρίζουν τις τροπολογίες μου. Στην περίπτωση αυτή είμαι ικανοποιημένη. Μάλιστα, ναι, ναι, είναι πολύ θετικό σημάδι, λέει η Πρόεδρος. Μάλιστα. Να σας πω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 6η Μαΐου, 17 η ώρα το απόγευμα, 5 η ώρα το α, απόγευμα. Θα ψηφίσουμε στις 30 Μαΐου και μετά στην Ανομέλεια 7, η Επιτροπή θα ψηφίσει 7 Ιουλίου.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 Ίσως θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε και ένα άλλο ε, σημείο, το οποίο έχουμε ε, προβλέψει για κάποια άλλη στιγμή στην ημερήσια διάταξη, ε, για την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών στις ΗΠΑ, που έλαβε χώρα πριν από δύο εβδομάδες. Αλλά δυστυχώς δεν έχω τα κατάλληλα έγγραφα μπροστά μου αυτή τη στιγμή, την έκθεση. ett ögonblick. Vi skulle inte ta den här punkten nu, så jag blev lite... Α, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα αυτό τώρα, δηλαδή. ja, då så. Ναι, λυπάμαι πάρα πολύ, ζητώ συγγνώμη. Αλλά δεν είχα υπολογίσει ότι θα ολοκληρώναμε τόσο γρήγορα την προηγούμενη ε, συζήτηση και δεν έχω μπροστά μου τα απαραίτητα έγγραφα. Αλλά από τις 2 μέχρι 4 Απριλίου μεταβήκαμε στα, ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ ως πρόεδρος ε, συμμετείχα και η κυρία Κράτσα συμμετείχε. Η κυρία Ροντζίλη από το ΕΛΚ και η κυρία Ολδέ από το ΑΛΔΕ. συμμετείχε και η γραμματεία και κάποια μέλη της Άλτα και φυσικά κάποιοι διερμηνείς προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και εύρυθμη λειτουργία. Την πρώτη ημέρα μεταβήκαμε στη Νέα Υόρκη, όπου συναντηθήκαμε με τη Μάργκο Βάλστρομ. η οποία ως αρμόδια επιτροπός για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρισκόταν εκεί. Συναντηθήκαμε και με διάφορους εκπροσώπους ε, οργανώσεων ή τα δικαιώματα των γυναικών. Η κυρία Πούλη, για παράδειγμα, και με άλλους εκπροσώπους ε, που για διάφορα θέματα, βία κατά των γυναικών, ε, ισότητα ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών στον εργασιακό χώρο, η συμπληρωμή γυναικών και ανδρών και νομίζω ότι το ενδιαφέρον που εκφράστηκε ήταν πραγματικά μεγάλο. Κάναμε πάρα πολλέ καλές επαφές από πλευρά τη Επιτροπή μας με τις ε, άλλες οργανώσεις και μετά ε, ταξιδέψαμε στην Ουάσιγκτον όπου συναντηθήκαμε με μία σειρά εκπροσώπων της κυβέρνησης, εκπροσώπους ε, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Εργασίας, συναντηθήκαμε και με μη κυβερνητικέ οργανώσει. επεξεργαστήκαμε τον τρόπο λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη ΣΥΠΑ σε ό,τι αφορά θέματα ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Ο πρόεδρος Ομπάμα το 2009 ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για την πρόθεση των δικαιωμάτων των γυναικών και αυτό αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο υποστηρίζει και η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Να ζητήσω από την κυρία Κράτσα ίσως να πει δύο λόγια. Αλλά γενικά νομίζω ότι μπορούμε να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι οι ΙΠΑ εν μέρη βρίσκονται λίγο πολύ στην ίδια κατάσταση που βρισκόμαστε κι εμείς. Ε, διαφορά μισθών, ε, προβλήματα βίας κατά των γυναικών. Όλα αυτά αποτελούν ζητήματα τα οποία θυμίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κι εμείς στη δική μας Ήπειρο. Προσωπικά θα πρέπει να πω ότι κατέληξα και σε ένα άλλο συμπέρασμα σε ό,τι αφορά την ε, κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Έχω την αίσθηση ότι οι γυναίκες στις Ήπα αντιμετωπίζουν πολύ πιο πολλά προβλήματα. Συχνά είναι πολύ πιο περιορισμένο το επίπεδο εκπαίδευση και κατάρτιση και πραγματικά χρειάζεται μεγάλη προσωπική επένδυση για την κατάρτισή τους σε κατάλληλες σχολές. Και νομίζω ότι υπάρχει έντονη η επιθυμία για πιο ε, εντατική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης και μεταξύ της Αμερικανικής κυβέρνησης και της Επιτροπής μας συγκεκριμένα. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας και πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε ε, εμπειρίες. Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατηρήση, αν μου επιτρέπετε. Φαίνεται επίσης Όταν συναντηθήκαμε με το White Council, ε, φάνηκε ξεκάθαρα πόσο υψηλό είναι το κύρος ε, που ε, έχει η Επιτροπή μας. η εκπρόσωπος του White Council καθυστέρησε λίγο στην άφηξή της και είχε συναντηθεί προηγουμένως με την πρώτη κυρία τον Ήπα μας ζήτησε πραγματικά ε, συγγνώμη και μετά από μία ώρα αναγκάστηκε να ξαναφύγει. Είχε άλλη συνάντηση με την πρώτη κυρία τον Ήπα αλλά ασφαλώς και ζήτησε συγγνώμη, αλλά να δώσω το λόγο στην κυρία Κράτσα για να μας αναφέρει τις δικές της εντυπώσεις. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να πω ότι η... θα ήθελα να πω λέω καταρχάς ότι η η πρωτοβουλία αυτή της επίσκεψης στις Ηνωμένες με το διπλό στόχο αφενός τους διεθνούς οργανισμούς και αφετέρου την ε, Αμερικανική κυβέρνηση ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Καταρχάς ε, ε, έδωσε μια ορατότητα και ενημέρωση προς την Αμερικανική και τη διεθνή πλευρά του ρόλου της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιο συγκεκριμένα της Επιτροπής μας, διότι επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι αισθανθήκαμε πρεσβευτές αυτού που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο του έργου της Επιτροπής μας. Ήθελα επίση να σας ευχαριστήσω για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο διευθύνατε αυτή την αποστολή και να ευχαριστήσω και τους, τα τους παρόντες ε, administrators της Επιτροπής μας για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο προετοίμασαν και μας συνόδευσαν σε όλη αυτή την αποστολή. Ε, συμφωνώ μαζί σας ότι διαπιστώσαμε ότι τα, το κοινωνικό ευρωπαϊκό κράτος, παρόλο τα, πλήγματα που έχει υποστεί λόγω της οικονομικής κρίσης, της δημοσιονομικής αστάθειας κτλ, κρατάει ακόμη γερά σε σύγκριση με το αμερικανικό. Αυτό ίσως δεν ήταν μια έκπληξη, ε, για μένα μια θετική έκπληξη είναι το πόσο στην Αμερική αναγνωρίζουν ότι εμείς έχουμε και ένα know-how ε, βαθύτερο και ευρύτερο από αυτό που έχουν οι Αμερικανοί. Σε κάθε επαφή μας αντιμετώπιζαν ως τους καλύτερα κρατούντες από ότι το αμερικανικό establishment. Ε, επίσης είδα ε, θετικά το ότι υπάρχουν οργανισμοί όπως δεν θυμάμαι ακριβώς το, το, Συμβούλιο των, Γυναικών στις Business που ήταν σε ένα ίδρυμα υποτροφιών του Πρόεδρου Γουίστον. Ε, ναι, ε, πόσο ενδιαφέρθηκαν ε, μου ξεφεύγει το όνομα, ενδιαφέρθηκαν να κρατήσουν την επαφή μαζί μας, διότι έχουν ένα πρόγραμμα ενημέρωσης γυναικών leaders, του τι είναι η Ευρώπη και πώς λειτουργεί. Πιστεύω ότι ε, υπάρχει ένα έδαφος πιο έφορο από αυτό που και εγώ με άλλες επαφές που είχα ήδη κάνει και με τους διεθνείς οργανισμούς και με την Αμερικανική κυβέρνηση, ε, πιο έφορο για διάλογο και προώθηση του ρόλου της Ευρώπης σήμερα. Πιστεύω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το, αυτό το περιβάλλον που δημιουργείται και μέσα από τον διατλαντικό διάλογο να βάλουμε, εγώ θα κάνω μια πρωτοβουλία και θα ήθελα να κάνω και μια έκθεση πρωτοβουλία αν το εγκρίνετε κύριε Πρόεδρε μαζί με τους συντονιστές για το ρόλο, το, για το, το gender θεμάτων στο πλαίσιο του διατλαντικού διαλόγου. Ε, πιστεύω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος, η παγκοσμιοποίηση γίνεται όλο και πιο έντονη, η, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, τους, κάνουν, τους φέρνουν όλο πιο κοντά για να υποστηρίξουμε το, το δυτικό μοντέλο του πολιτισμού, ε, την οικονομική ανάπτυξη, όλα αυτά είναι θέματα, η συμμαχία μας στο G20, στο G8, όλα αυτά είναι θέματα που μας φέρουν πιο κοντά και φέρνουν τη γυναικεία διάσταση της προσπάθειάς μας πιο έντονη και πιστεύω ότι πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Δεύτερον, και συγγνώμη θα φύγω γιατί έχω ένα ραντεβού με τον γιατρό, ε, δεύτερον ο, ο, ήθελα να πω και στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών εντυπωσιάστηκα το πόσο ήταν προετοιμασμένοι ακόμη και για την ατζέντα μας. Ε, τα θέματα που έχουμε να συγηθούμε ε, και τα οποία άπτονται της αναπτυξιακής βοήθειας. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κρατήσουμε την επαφή ε, και να επαναλάβουμε αυτή την επίσκεψη με μια άλλη ευκαιρία, διότι είναι προ όφελο των αξιών και των πολιτικών που υπηρετούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει σχόλια να κάνετε να αρχίσουμε την συζήτηση. Η κυρία Γκουρμά έχει το λόγο. Συμμετείχα και εγώ στην αντιπροσωπεία. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να μεταβώ. Ε, δεν μπόρεσα να συμμετέχω στις ψηφοφορίες, γιατί έπρεπε να συμμετάσχω σε άλλες ψηφοφορίες, σε άλλη επιτροπή, όπου μετρούσε και τελευταία ψήφος. Αλλά να πω ότι υποστηρίξω, να πω ότι υποστηρίζω την ε, θέση σας και είναι σαφές ότι εφόσον έχουμε και γραφείο στην Ουάσιγκτον, είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθεί τις ιδέες αυτές με το σωστό τρόπο. Θα ήταν πάρα πολύ καλό αν ο κύριος Φεσλέγγιν είχε επισκεφτεί την ε, η κυρία Χουσλέγκερ μάλλον είχε επισκεφθεί το κοινοβούλιο και την επιτροπή μας μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκε το κοινοβούλιο. Καλό θα ήταν όμως να γίνει και άλλη μια συζήτηση στην επιτροπή τη δική μας. Κάποια στιγμή το φθινόπωρο αν θα μπορούσατε να, την ε, καλέσετε. Νομίζω ότι θα είναι καλό να συζητήσουμε και τους στόχους της χιλιετίας και πολλά άλλα. Και είχα ταξιδέψει στις ΗΠΑ πριν από ένα μήνα και συναντήθηκα με πολλούς αρμόδιους και μας είπαν ότι πραγματικά θέλουν να ξεκινήσουν δράσεις ε, από κοινού μαζί μας, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό. Θα ήταν πάρα πολύ θετικό λοιπόν να έρθει να μας επισκεφθεί και να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε και πόσο μπορούμε να συνεργαστούμε. Μου προκάλεσε λοιπόν κάποια απογοήτευση το γεγονός ότι δεν μπορέσα να συμμετάσχω και εγώ στην αποστολή, αλλά επειδή είναι η τελευταία ημέρα σας ε, ως πρόεδρος, να σας πω ότι είναι κρίμα που φεύγετε, ήταν εξαιρετική η συνεργασία. Ελπίζω να μείνετε παρόλα αυτά μαζί μας και να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Εγώ Ήμουν τυχερή γιατί σας ήξερα και από άλλες επιτροπές. Ξέρω ότι είσαστε πάρα πολύ δεσμευμένοι, νεαρή γυναίκα, με πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό. Ελπίζω να βρείτε λοιπόν μια καλή θέση και ελπίζω ότι ο πρόεδρος θα σας υποστηρίξει και αυτός. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Επομένως, να σας πω το εξής. Αν καταρτήσουμε κάποια έκθεση γνωμοδότηση, φυσικά αυτό θα συζητηθεί στο μέλλον, θα είναι αντικείμενο του επόμενου προγράμματο εργασία μα. Τώρα, κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να καταρτήσουμε μια επιστολή, να συντάξουμε μια επιστολή και να τη στείλουμε στον πρόεδρο τη ε, ε, αμερικανικής αντιπροσωπείας, στο Κοινοβούλιο για την Αμερική και να πούμε ότι η Επιτροπή μας επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και να συντάξουμε μια έκθεση της επισκεψής μας και αυτός είναι ένα τρόπος να ενημερώσουμε για την επίσκεψή μας ε, τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ελευθέντως αυτού. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη και Έχουμε κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας, γιατί η Επιτροπός Ρέντινγκ θα έλθει στις 10.30. Θα αναστείλουμε λοιπόν τώρα τη συνεδρία, θα διακόψουμε και θα επανέλθουμε στις 10.30. Okay, welcome everybody. Uh, I'm gonna swap. Καλώς ήρθατε και θα μιλήσω Σου σουηδικά. Για βάλτε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Είναι τόσο καθαρά τα σουηδικά μου, τα καταλαβαίνετε και χωρί ακουστικά σα κατάλαβα. Καλώ ήρθατε όλοι λοιπόν εδώ. Ιδιαίτερα δε καλωσορίζω εσά. Κυρία Ρέντα, κυρία Επίτροπε, χαίρομαι ιδιαίτερω που σας βλέπω εδώ σήμερα και αυτή την ανταλλαγή απόψεων και στενό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδιαίτερος χαίρομαι για την ύπαρξη μέτρων από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια νέα δέσμη προτάσεων που μας αποσχολεί και εμάς που μπορεί να αποτελέσει μια καλή λύση, πιστεύουμε, σε συνεργασία και με το Συμβούλιο, μέσα από τι διαπραγματεύσει, που τη σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για του πολύ σημαντικού στόχου που έχουν προσδιοριστεί στην ε, προοπτική ιδιαίτερω ε, την σχετική με το φύλλο που μας ενδιαφέρει Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που ήρθατε σήμερα. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε ό,τι έχετε να μας πείτε. Υπάρχουν διάφοροι τομείς, όπως η παραδείγματι η βία που προσανατολίζεται στο φύλλο. Ή θέματα που βάζουμε και στις προτάσεις σας, δηλαδή καλύτερο συγκερασμό του οικογενειακού και του ε, επαγγελματικού βίου, που μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα θέμα το οποίο είδαμε και στην ψηφοφορία μας με μια πολύ σημαντική έκθεση. Ισότιμη αμοιβή για ίση αξίας εργασία. Είναι ένα άλλο θέμα στο οποίο χρειάζεται να κάνουμε περισσότερε προσπάθειες. Δεν, δεν έχει προχωρήσει αρκετά η υπόθεση αυτή εδώ και πολύ καιρό έχει μείνει η νομοθεσία, η ενισχύει και πρέπει να αναλάβει κάποια δράση. Η Επιτροπή πιστεύω διότι μπορεί να αποτελέσει η διαφορετική αμοιβή ε, και λόγω διάκρισης εις βάρος των γυναικών και άρα μεγάλες διαφορές σε επίπεδο αμοιβών να ε, θέσουν σε δυσμενέστερη και κοινωνικά θέση της γυναίκες γενικότερα, φέρει πίνος προς την ε, εξασφάλιση ταξιδοτικών δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Πάντως χαιρόμαστε πολύ σας βλέπουμε εδώ και περιμένουμε με να ακούσουμε τις προτάσεις σας. Η κυρία Ρέντινγκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζετε ασφαλώς από την εμπειρία σας ότι αυτός ο διαρθρωμένος διάλογος αποτελεί μια ευκαιρία για να ε, καταγράψουμε τι εξελίξει σε μια ε, υπόθεση, σε διάφορα θέματα ε, και να προτείνουμε νέους δρόμους πρόοδου. ιδιαίτερο εκτιμώ τι προτάσεις και τις προσπάθειες της Επιτροπής σας ε, στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αναφερθώ σε διάφορα θέματα. Καταρχάς τα θύματα. Εκφράσατε ισχυρή υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις που εξελίσσονται σε σχέση με την οδηγία για ελάχιστα δικαιώματα των ε, θυμάτων. Τη σημαντική αυτή έκθεση την ψηφίσατε εκθέση Παρμάνοβα και Χιμένες Μπεσερίλ. Ε, πρόοδο επίση σημειώσατε στο τριμερή διάλογο. Και έτσι πιστεύω ότι σε συνεργασία και με τις συγκεκριτές μπορούμε να έχουμε πολύ καλή και ισορροπημένη πρόταση. Θα ήθελα να ευχαριστώ εσάς το Κοινοβούλιο, διότι ιδιαίτερη έμφαση δώσατε στα θύματα της βίας που σχετίζεται ή αναφέρεται στο φύλλο. Μέσα από την έκθεση αυτή. Πρόκειται για μια προσέγγιση την οποία και εγώ ε, ε την οποία και εγώ παρακολουθώ ιδιαίτερως. Επίσης, Έχουμε, σε σχέση με την προστασία των θυμάτων, την, την πρόοδο ήδη καταγεγραμμένη στο ποινικά ζητήματα. Τώρα μας έχει μείνει η αστική πτυχή. Ξέρετε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν, ε, έχουν καθεστώς προστασίας θυμάτων για την ποινική δικαιοσύνη αλλά έχουν και στην αστική αλλά και στη διοικητική ακόμη δικαιοσύνη ε, καθεστώ προστασία θυμάτων. Έτσι εξασφαλίζεται μια πλήρη ομπρέλα κάλυψη των θυμάτων και γι' αυτό πρέπει να επεκταθεί αυτό το σύστημα και ε, πέραν της ποινική και στην αστική δικαιοσύνη. Γι' αυτό αισθάνομαι ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την ε, εισηγήτρια κυρία Παβάνοβα για την ιδιαίτερη στράτευσή της, τις προσπάθειές της και το εργαστήριο συστήσεων που οργάνωσε πρόσφατα στην Επιτροπή σας. Πολύ σημαντικό διότι πρέπει να αντιληφθούμε πώς ε, διαφορετικά μέτρα αναπτύσσονται σε διαφορετικά κράτη-μέλη και πώς ε, πρέπει να συνεργαστούμε για να ε, αναπτύξουμε τα μέτρα αυτά. Γιατί μια γυναίκα σε κίνδυνο δεν ε, έχει την πολυτέλεια να εξετάσει τις λεπτομέρειες της κάθε εθνικής νομοθεσίας, θέλει απλώς ταχύτατα να της προσφερθεί η προστασία. Γι' αυτό λοιπόν ε, ιδιαίτερα ευγνωμονούμε για την οργάνωση του εργαστηρίου συζητήσεων που μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την νομοθεσία ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες για προστασία το ζήτημα της ε, κλειτοριδεκτομής. Επίσης, θα ήθελα να σας αναφέρω εδώ ότι προσφέρεται και και οικονομική στήριξη για την εφαρμογή ε, διεθνικών ή πολυεθνικών προγραμμάτων ε, για την αντιμετώπιση αυτών των πρακτικών της κλειτοριδεκτομής. έχουμε ζητήσει μια μελέτη για καταγραφή της κατάστασης και των τάσεων στο πρόβλημα αυτό, γιατί ξέρετε έχουμε μόνο εμπειρική γνώση περιστασιακή, κατακαιρματισμένη, που κυρίως μας προσφέρουν οι κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται στην υπόθεση αυτή, ε, χωρίς όμως να έχουμε μια ουσιαστική χαρτογράφηση της κατάστασης. Αυτό λοιπόν είναι το αντικείμενο των εργασιών της Ομάδας Εργασίας για την Ισότητα που ε, έχει αναλάβει το καθήκον της χαρτογράφησης και θα υποβάλει τη σχετική της έκθεση το 2012 βάσει της οποίας στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και θα λάβουμε αποφάσεις για το πώς μπορούμε να δράσουμε για να καταπολεμήσουμε αυτή τη μορφή της βίας εις βάρος νεαρών κοριτσιών που είναι απαράδεκτη. γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια. Ξέρετε ότι οι γυναίκε σε, ε, σε υψηλές θέσεις αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων είναι ένα θέμα που επίση μα ενδιαφέρει πολύ και που αποτελεί προτεραιότητά μας. Ε, βάση και επιστημονικών στοιχείων γνωρίζουμε ότι η ισότητα των φύλων εξασφαλίζει η οικονομική ανάπτυξη και άρα υπάρχουν και σημαντικά οικονομικά επιχείρημα για την ε, συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και κυρίως στις θέσεις ε, αρμοδιότητας ε, ανά την Ευρώπη. Άρα αυτό είναι ένα αποδεδειγμένο επιχείρημα, το ότι πρέπει δηλαδή να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των γυναικών στις ε, θέσεις των στελεχών, ε, στις αποφάσεις. Ε, το θέμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι το πώς θα τα καταφέρουμε. Στηριζόμαστε στις προτάσεις της κυρίας Κράτσα του 2011. Η κυρία Νατφέλ και η κυρία είναι φέτος ανέλαβαν αυτό το καθήκον και έχετε στήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις νομοθετικέ Εγώ παρακολουθώντας ε, τις ε, συζητήσεις σας και τις προτάσεις σας, ανέλαβα την πρωτοβουλία για δημόσιο διάλογο, πολύ συγκεκριμένο, όχι απλώς δηλαδή γενικόλογη συζήτηση για το πώς ή το εάν, μια, ένα δημόσιο διάλογο ο οποίος ε, θα συνεχίσει για αρκετό καιρό για να εντοπιστούν τα συγκεκριμένα προβλήματα και οι λύσεις. Στη συνέχεια θα ε, αναλάβω συστήσεις με τους συναδέλφους στην Επιτροπή για να δούμε πώς περαιτέρω θα ε, αντιμετωπίσουμε το ζήτημα στο υπόλοιπο του έτους. Το ζήτημα της οδηγίας και την αδιαμετρότητα. Για να ε, αρκετά συναισθήματα δυσφορίας και ματέωσης. Είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω στο οποίο πιστεύω πολύ περιμένουν πρόοδο. Έχω εργαστεί σε στενή συνεργασία με τις τρεις τελευταίες προεδρίες, προεδρίες για να ενθαρρύνω την πρόοδο στην υπόθεση αυτή. Πρέπει να πω ότι... Θα ήθελα να τονίσω ότι η Πολωνική Προεδρία οργάνωσε ειδικέ συναντήσεις των Υπουργών μόνο για τα θέματα αυτά της ημερήσιας διάταξης και νομίζω ότι όλα Όσα μπορούσαν να γίνουν έγιναν. Και πρότεινα στους υπουργούς την ιδέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ιδέα της ρήτρας Πασαρέλ, που θα επιτρέπει διάφορες προβλέψεις σε διάφορα την αδιαμετρότητα και η Ιδανική Προεδρία κινείται προς την κατεύθυνση αυτή και η Κομισιόν θα κάνει όλες τις προσπάθειες που μπορεί να υποστηρίξει την πρωτοβουλία αυτή. Τούτου λεχθέντος, θεωρώ ότι στην ε, παρούσα φάση είναι ελάχιστη προσπάθεια που καταβάλει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω, να μου πείτε, τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση για το πρόβλημα αυτό, δεδομένου του ότι όλες οι προσπάθειες που έχω καταβάλει δεν έχουν ε, ε, καρποφορήσει σε ό,τι αφορά την άρση των φραγμών. Μία άλλη ιστορία η οποία επίσης δεν έχει ε, στεφτεί με επιτυχία η οδηγία του άρθρου 19 για την ίση αντιμετώπιση μπλοκάρεται από πολιτική αντίσταση κάποιων κρατών μελών, παρά το γεγονός ότι υπάρχει πλειοψηφία υπέρ της οδηγίας στο Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι εκφράζονται ανησυχίες για συγκεκριμένες πτυχές, αυτό όμως είναι κάτι που μπορεί να επιληθεί ασφαλώ. Η οδηγία ωστόσο προαπαιτεί ομοφωνία. Εδώ και κάποια χρόνια λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το σχέδιο οδηγίας, υποστηρίζει όλες τις προεδρίες που συνέρχονται σε τεχνικές συναντήσεις για την οδηγία αυτή Όλα αυτά καλά και ωραία, αλλά επιμένει η πολιτική αντίσταση. η διαφορά μισθολογική μεταξύ των φύλων. Ξέρετε ότι αυτό αποτελεί τμήμα της ε, στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική για το 2010-2015. Και ξέρετε ότι ο ίσος μισθός καταχωρίζεται, κατοχυρώνεται και στις ε, σχετικές συνθήκες. Ξέρετε ποια είναι τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία. Ξέρετε ότι υπάρχει μείωση από το 17,6% στο 16,4% κατά μέσο όρο, σε ό,τι αφορά το χάσμα δηλαδή, αλλά σε κάποιες χώρες ε, οι διαφορές αυτές ε, οξύνονται. Θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι το πρόβλημα αυτό είναι πολύ σύνθετο και έχει πολλές, πολλαπλές αιτίες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι γενικά οι άντρε βγάζουν πιο πολλά από ότι οι γυναίκε, θα πρέπει να εξετάσουμε και τις βαθύτερε αιτίε πίσω από το φαινόμενο αυτό και θα πρέπει να είναι πολλαπλών επιπέδων οι προσεγγίσεις μας. Και θα πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία και με τα θεσμικά όργανα και με τα κρατή μέλη, με τα συνδικάτα και με τις ενώσεις εργοδοτών. Το καλό έργο της κυρίας ε, εισηγήτριας Μπάουερ απέστειλε τα σωστά μηνύματα προς την κατεύθυνση αυτή. Καταρχάς, θα πρέπει να εφαρμόσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία, τους υφιστάμενους κανονισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θέματοφύλακας των συνθήκων το πράττει αυτό. Καταχωρούμε, ε, ε, ε, εξετάζουμε και παρακολουθούμε που εφαρμόζονται σωστά και που όχι οι φυστάμενες νομοθεσίες και το 2013 θα α, δημοσιευθεί σχετική έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας. Κατά δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντική η ευαισθητοποίηση για να είναι όλοι ενήμεροι για το γεγονός ότι το θέμα αυτό μας ανησυχεί, εξακολουθεί να μας ανησυχεί, δεν το έχουμε ξεχάσει. Να θυμάστε ότι η δεύτερη ημέρα για την ε, ίση ε, μισθολογική ανταμοιβή ήταν η 2η Μαρτίου και διοργανώθηκαν διάφορες ε, ε, εκδηλώσεις που τόνιζαν ακριβώς το πόσο παράλογο είναι να υπάρχει τέτοιο χάσμα μεταξύ των μισθών των γυναικών και των ανδρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσης μια πρωτοβουλία για να ευαισθητοποιήσει και τις επιχειρήσεις, τις εταιρείε. Θα προωθήσει ε, εκπαιδευτικές δραστηριότητες ε, σε ό,τι αφορά το σκέλος το επιχειρηματικό για την ισότητα των φύλων. Συνεργάστηκα επίσης με οργανώσεις του οικονομικού κλάδου, του βιομηχανικού κλάδου, προκειμένου σωστά να ενημερώσουν τα μέλη τους για το τι συμβαίνει. Και αυτό με οδηγεί λοιπόν στο τρίτο στοιχείο, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τη, τους μισθούς. Στο σημείο αυτό ακολουθούμε τις δράσεις, τα πιλωτικά προγράμματα στην Πορτογαλία, στη Γερμανία και στην Αυστρία που έχουν εφαρμόσει σχετικά μέσα σε ό,τι αφορά την διαφάνεια. Παρακολουθούμε λοιπόν πώς εξελίσσονται αυτά τα μέσα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους. Ένα άλλο σημείο, Πρόεδρε, το οποίο θα γνωρίζετε. Υπάρχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θα γνωρίζετε όμως και ότι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτό όλα τα κράτη-μέλη καλούνται να παρουσιάσουν τις εθνικές τους στρατηγικές. Όλα λοιπόν τα κράτη-μέλη όντως παρουσίασαν τις εθνικές τους στρατηγικές και πραγματικά δεν ήταν εύκολο το εγχείρημα, τα καταφέραμε όμως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη φάση ανάλυσης και αξιολόγησης των εθνικών αυτών εκθέσεων, θα δημοσιευτούν τα σχετικά αποτελέσματα σύντομα. Και επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι το νέο πρόγραμμα για τα δικαιώματα των πολιτών θα συμπεριλάβει και το θέμα της ε, ε, ένταξης των Ρωμά μεταξύ των προτεραιοτήτων γιατί δεν ήταν προτεραιότητα στο Solvit. Τι θέματα προσβασιμότητας. Θα σας ε, ενδιαφέρει να ακούσετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει ένα σχέδιο, μια πράξη ευρωπαϊκής προσβασιμότητας προκειμένου να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή αγορά των προσβάσιμων υπηρεσιών και προϊόντων όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους ανάπηρους αλλά και για τους ηλικιωμένους όσο γυράσκουν τόσο αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας. Τέτοιες λοιπόν προϋποθέσεις ε, προσβασιμότητας ε, καταργώντας εμπόδια μεταξύ της ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών μελών λόγω των ε, διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών. Θα είναι διτό το έργο μας, θεωρώ, ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε ένα προσβάσιμο περιβάλλον στους ανάπηρους και στους ηλικιωμένους και παράλληλα να σπρώξουμε, να δώσουμε κίνητρα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, στον ευρωπαϊκό οικονομικό κλάδο, προκειμένου να δημιουργηθούν τα αγαθά και υπηρεσίε που χρειάζονται για τα άτομα αυτά. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο θέμα δικαιωμάτων, αλλά και θέμα ανάπτυξη, αν θέλετε. Και τέλο, το τελευταίο ζήτημα που ήθελα να σα αναφέρω. Αυτή αένα η ιστορία με την γραμμή έκτακτης ανάγκης για τα παιδιά τα αγνοούμενα παιδιά. Μια ευρωπαϊκή γραμμή για την αναφορά αγνοούμενων παιδιών. Προσπαθούμε να πιέσουμε τα κρατη προκειμένου να καταστεί λειτουργική η γραμμή που ήδη είναι λειτουργική σε 17 ε, κρατημέλη, αλλά όχι και στα 27, δυστυχώς ακόμα. Θα συνεχίσω να καλώ τα κρατημέλη να εφαρμόσουν αυτή τη γραμμή την τηλεφωνική για τα αγνοούμενα παιδιά το συντομότερο δυνατόν και καλώ όλους τους εμπλεκόμενους ε, φορείς, τα κράτη-μέλη, τους εθνικούς ρυθμιστικούς ε, φορείς, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ούτω καθεξής να συνεργαστούν. Θα διοργανωθεί ένα συνέδριο τέλη Μαΐου που και πάλι θα φέρει σε επαφή όλους τους φορείς αυτούς και ασφαλώς και θα είναι προσκεκλημένο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο συνέδριο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ήταν να ακούσουμε το πρόγραμμα της Επιτροπής. Και τώρα ήρθε το πληρωματικό να ακούσουμε τους βουλευτές. Αλλά θα δώσω καταρχήν το λόγο στην κυρία Χάνιμπολ που είναι η εισηγήτρια για θέματα προπολογισμού. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο. Ήταν πολύ περιεκτική η δήλωσή σας και όλοι ξέρουμε ότι ε, δίνετε πολύ μεγάλη σημασία σε θέματα που αφορούν τη ισότητα των δύο φίλων. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας και για την τεράστια δουλειά που έχετε κάνει από αυτού. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω κάποια θέματα με τη σειρά και θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα της βίας κατά των γυναικών με το οποίο ασχολούμαστε σε αυτήν την Επιτροπή για πάρα πολύ καιρό όπως, όπως γνωρίζετε και η βία ε, αυτού του είδους, ε, λόγω του φύλου δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντική και δυστυχώς δεν εξαφανίζεται. Έχουμε δεσμευτεί ε, για την καταπολέμηση αυτής της βίας εδώ και καιρό και ξέρουμε τα όσα κάνατε και ζητάμε εδώ και κάποια χρόνια για μια πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών για μια συνολική στρατηγική. Ξέρω ότι εργάζεστε Γι' αυτό το θέμα και οι δέσμοι μέτρων για την προστασία των θυμάτων ε, είναι ένα καλό βήμα, αλλά θέλουμε μια συνολική στρατηγική, όπως αναφερόταν και στο πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμη. Αυτό θα είναι βασική προτεραιότητα για μας, για την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών ε, και για φέτο και για το πρόγραμμα του 2013. Και με αυτό το θέμα συνδέεται το ζήτημα της κλητροδοκτομής που δείξατε κι εσείς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι συνεχίζονται οι εργασίες στον τομέα αυτό και ότι ε, γίνεται έρευνα υψηλής ποιότητας και υπάρχει υποστήριξη για διεθνικά προγράμματα. Θέλω να τονίσω επίσης ότι πάρα πολλά λαμβάνουν χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σύμφωνα, είχαμε μάλλον μία πρόσφατη έκθεση που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και εγώ εκπροσωπώ το Λονδίνο όπως γνωρίζετε και είναι μεγάλο αυτό το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και εντός των συνόρων μας όπως και στο υπόλοιπο κόσμο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, αυτό το θέμα, είναι κρυφό και πάρα πολλές φορές δεν είναι εμφανές το πρόβλημα αυτό στις κοινότητες, στα κράτη-μέλη μας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας ε, και να το επεκτείνουμε έτσι ώστε να περιλάβουμε όλα τα θύματα. Θα ήθελα να αναφέρω και το πρόγραμμα Δάφνη, το οποίο όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε και όλοι μας ήταν ε, πάρα πολύ καλό, σημείωσε τεράστια επιτυχία και ελπίζω να έχουμε μία διαβεβαίωση ότι θα προστατευτεί το πρόγραμμα Δάφνη από τις περικοπές του προπολογισμού. Ξέρω ότι υπήρξαν απειλές ε, κατά του προγράμματος ε, και θέλω να σας παροτρύνω να διασφαλίσετε ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα Δάφνη, θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται στα σημερινά επίπεδα, αν όχι περισσότερο, γιατί έχει πάρα πολύ καλή φήμη και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Να προχωρήσω τώρα στο θέμα της ε, λήψης αποφάσεων, ε, πόσο οι γυναίκες συμμετέχουν στη λήψη, στη λήψη αποφάσεων. Ξέρω ότι υπήρξε ευαισθητοποίηση για το θέμα αυτό και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν ε, ανακοινώσατε αυτή την πρωτοβουλία στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, όλα τα μέσα ενημέρωση αναφέρθηκαν σε αυτό και όχι με εχθρικό τρόπο, μάλιστα με αρκετά ενθαρρυντικό τρόπο. Η σημερινή κατάσταση θεωρηθήκε ότι δεν είναι αρκετά καλή και οι περισσότεροι σχολιαστές ε, εκτός ίσως από την κυβέρνηση, αλλά όλοι οι υπόλοιποι θεώρησαν ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Αυτό είναι εξαιρετικό και πραγματικά ε, νομίζω ότι εδώ ε, δεν χρειάζεται να επιμείνουμε, είναι όλοι πεισμένοι, αλλά ξέρω ότι θα συνεχίσετε την καλή δουλειά και θα σας υποστηρίξει και η Επιτροπή μας. Επίσης, ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι συμμετέχουν περισσότερες ε, γυναίκες στην ε, λήψη πολιτικών αποφάσεων. Βελτιώνεται η κατάσταση, αλλά σε ορισμένα κρατημέλη δεν είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι και εμείς πρέπει να το πράττουμε αυτό ως Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών σε ένα εκλεγμένο όργανο. Θα ήθελα να δω εμείς να κάνουμε περισσότερα, να διατηρήσουμε την ορμή και να οθήσουμε τα κράτη-μέλη στο να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες ε, στη ε, συστήματα τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και στην κατάρτιση της νομοθεσίας. Στα σχέση με τα άλλα θέματα που θίξατε, θα ήθελα φυσικά να αναφερθώ και εγώ στο μισθολογικό χάσμα. Ε, ψηφίσαμε αυτή την έκθεση σήμερα το πρωί. Έχουμε τώρα ένα σχέδιο οδηγία ε, από αυτή την Επιτροπή και θέλουμε να ελεγχιστοποιήσουμε αυτό το μισθολογικό χάσμα. Εργαζόμαστε πολύ καιρό στο θέμα αυτό και θέλω να συνεχιστεί και σε συνεργασία με την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι αμοιβοί που λαμβάνουν οι γυναίκε είναι η ίδια και να τεθεί τέλο σε αυτή την αδικία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχει ανισότητα τη αμοιβή. Είναι πολύ πλοκό το πρόβλημα, όπω είπατε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες ε, αμείβονται το ίδιο. Και όπως είπατε, δεν υπάρχει διαφάνεια στους μισθούς ε, και ε, πάρα πολλά πράγματα από τα οποία μιλάμε στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών, αν και ωφελούν τις γυναίκες και γι' αυτό τα κάνουμε, επίσης ωφελούν και την κοινωνία συνολικά και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, ε, πολλέ φορέ βελτιώνοντα τη θέση των γυναικών, βελτιώνουμε στην πραγματικότητα και τη θέση των ανδρών και όλη τη κοινωνική δομής και βελτιώνουμε την καθημερινότητά μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί και εμείς σε αυτή την Επιτροπή εδώ και πολύ καιρό ασχολούμαστε με το να θέσουμε τέλος στο Μεστολογικό κάσμα. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό που άκουσα για τους Ρωμά. Θα ήθελα αυτή η πρωτοβουλία να ανοίξει για να συμπεριλάβει και άλλες εθνοτικές ομάδες. Δηλαδή αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολλές άλλες ε, χώρες, ε, σε πολλές άλλες χώρες έχουμε ανθρώπους που έρχονται από άλλα μέρη του κόσμου και υπάρχουν ε, πολύ συχνά εντάσεις και δυσκολίες στο πώς αυτές οι κοινότητες συμβιώνουν με τους υπόλοιπους πολίτες. Έτσι λοιπόν, ε, νομίζω ότι είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία για τους Ρωμά, αλλά θα ήθελα να επεκταθεί για να συμπεριληφθούν και άλλες ε, κοινότητε εθνοτικών μειονοτήτων. Και θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας το θέμα τη ε, άδεια πατρότητα. Ξέρω ότι αναφέρατε την αδιαμητρότητα και ήταν βήμα τη οδηγία για την αδιαμητρότητα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω πού βρισκόμαστε σε σχέση με το θέμα της άδεια πατρότητα. Αυτά τα θέματα ήθελα να θίξω εγώ και σας ευχαριστώ για την συλλογική σας τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους ευρωβουλευτές. Πολλοί θέλουν να πάρουν το λόγο γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Επίτροπο. Θα πρέπει να περιορίσουμε το χρόνο ομιλία. Οι συντονιστέ θα έχουν δύο λεπτά στη διάθεσή του ο καθένα, γιατί θέλω να έχει και η Επίτροπο την ευκαιρία να απαντήσει τι ερωτήσει σα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους συντονιστές και θα ακολουθήσουμε τη σειρά του μεγέθους των ομάδων και κατόπιν τα υπόλοιπα μέλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερος ε, για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερος για τόσο πλούσια παρουσίαση και ιδιαίτερος για την δουλειά που έχετε μέχρι τώρα κάνει. Πάντοτε μπορείτε να στηρίξετε στην, υποστήριξη της Επιτροπής μας. Ερωτήσεις ε, για τη βία εις βάρος των γυναικών. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία σήμερα. Το πρόβλημα είναι η συγκρισιμότητα και η πρόσβασιμότητα στα δεδομένα αυτά. Ρωτώ λοιπόν τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να να βελτιστοποιήσει την ε, δική της συμβολή στην αντιμετώπιση του ζητήματος ε, και βέβαια πρέπει να πω ότι είχαμε μια πολύ καλή ε, ανταλλαγή απόψεων με την Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την ισότητα των, και τον, την οργάνωση για την ισότητα των φύλων και θα ήθελα να μας πείτε κάποιε συγκεκριμένε προτάσει για τι γυναίκε στα διοικητικά συμβούλια, στι ηγετικέ θέσει. Ε, θα πρέπει να συνεχίσει η διαβούλευση, όπω είπατε, και το Μάιο. Ωραία, ε, σε επίπεδο κρατών μελών πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια δημοσίευση των αποτελεσμάτων που θα ε, ε, μεταφραστεί σε λήψη νομοθετικών μέστρων. Τρίτη ερώτηση, ε, μισθολογικέ αποκλήσει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και πάλι με ενδιαφέρει να έχουμε δεδομένα που θα, θα είναι δυνατόν να μην δημοσιευθούν το 2013. Και ρωτώ πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια προσβασιμότητα πρόσβαση στι πληροφορίε και δεδομένου δε ότι οι επιχειρήσει δεν είναι καν υποχρεωμένε να μα δώσουν στοιχεία. Στην έκθεση τη κυρία Μπάουερ επίση θα ήθελα να μάθω ποια είναι η συνέχεια που σκοπεύετε να δώσετε σε μία από τις προτάσεις δυνατότητα, δηλαδή για να αναθεώρηση το άρθρο 20 της ε, Οδηγίας 2654, η οποία ε, προβλέπει την ενίσχυση των ε, της ισχύως της παρουσίας των γυναικών και άρα και τη μείωση των μισθολογικών αποκλήσεων. Επίσης, ε, για το έτος της Ιθαγένειας, το 2010, επεσήμανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγάλο εμπόδιο ως προς την Ιθαγένεια. Ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητες, στις οποίες εσείς θα επικεντρωθείτε για να δώσετε απαντήσεις και λύσεις το 2013. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόμψεν, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και εγώ από πλευρά μου. Ήταν πολύ διεξοδική η παρουσία σας κυρία Επίτροπε. Είμαι πιο αισιόδοξη πρέπει να πω. Και με ένα παράδειγμα θα το εξηγήσω ότι με προσκάλεσαν σε μία διημερίδα ε, για σχετικά θέματα στην οποία μιλούν ε, από 29 ομιλητές, 29 άντρες, ούτε μία γυναίκα δηλαδή δεν φαίνεται να συμμετέχει στην ημερίδα αυτή, να είναι προσκεκλημένη για να ομιλήσει επισήμω. Ε, άρα ε, μπορεί να είμαι εγώ αισιόδοξη, αλλά γενικώ η κατάσταση είναι μάλλον αρνητική και βλέπουμε ότι υποβαθμίζεται όλες τι βάρο των γυναικών. Ε, έχετε κάποιες προτάσει να μας δώσετε και τι ξέρω ότι δεν έχετε τελειώσει τη δουλειά σας αυτή. Περιμένουμε όμως. Περιμένουμε να δούμε και ποια είναι η θέση των κράτων μελών. Σε μια περίοδο δέο που τα κράτη-μέλη ασχολούνται με την οικονομική κρίση παρά με την ισότητα των φύλων, πρέπει εμείς να επιμένουμε ιδιαίτερως. Επίσης για τη διαφάνεια και τις μισολογικές αποκλήσεις πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερως ε, και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουμε πολλές ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 90% των γυναικών στη δική μου πατρίδα παραδείγματι απασχολούνται σε μικρές επιχειρήσεις με εργαζόμενους λιγότερους από 30, από 35. Γι' αυτό λοιπόν, εάν πούμε, ε, αν ορίσουμε ένα ποσοστό εργαζομένων, έναν αριθμό εργαζομένων ε, πολύ υψηλό, όπως προφτύρεται στην ε, οδηγία, τότε θα έχουμε πολύ περιορισμένη κάλυψη αυτού της μισθολογικής αποκλήσεως. Μην ξεχνάμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρώπης, άρα θα πρέπει να ορίσουμε για να είναι διαφανής διαδικασία ω ελάχιστο, ως ελάχιστο αριθμό εργαζομένων τους 10. Κυρία Παρβάνοβα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την παρουσία σας και την έκθεσή σας. Εκτιμούμε ιδιαίτερο στην ε, σταθερότητα με την οποία έρχεσαι στην Επιτροπή μας. Μας ε, μιλάτε με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Σημειώνουμε την πολύ καλή συνεργασία μαζί σας. Σημειώνεται επίσης και πολύ καλή πρόοδος χάρη στη συνεργασία αυτή. Και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσωπική σας στράτευση τον προσωπικό σας αγώνα και την υποστήριξη στην ομάδα του τριμερούς διαλόγου για την οδηγία. Φαντάζομαι ότι και για την προστασία των ε, θυμάτων στις αστικές υποθέσεις το ίδιο θα συμβεί και πάλι. Προσπαθούμε σε συνεργασία και με τους δικούς σας εμπειρογνώμους από την Επιτροπή να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή προστασία όχι μόνο με γνώμονα την ισότητα, αλλά και για να παρουσιάσουμε τις ιδέες μας και να εξασφαλίσουμε καλύτερη προστασία των θυμάτων και κυρίως αυτών που πέφτουν θύματα της προσανατολισμένης στο φύλλο βίας. Και θέλουμε τα θύματα να τα κοιτάζουμε μεμονωμένα σαν πρόσωπα και όχι ουδέτερα και απρόσωπα σαν ένα φάκελο μόνο που περνάει μέσα από το σύστημα για επεξεργασία. Εγώ το του λοιπόν θα θέλω να πω ότι η ε, κάθε προσπάθεια και με κυβερνητικέ οργανώσει, η εμπλοκή αυτών και καθενό θα πρέπει να στηριχθεί από εσά, αλλά και δημοσιονομικά, όχι μόνο ηθικά. Η δημοσιονομική λοιπόν υποστήριξη, η οικονομική υποστήριξη προ τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, ώστε να τις στηρίξουμε στη συνεργασία του με τι ή στι σχέσει του με τις εθνικές αρχές Γιατί πρέπει να αναπτύξουν τι δραστηριότητε εκείνες που θα τις επιτρέπει, θα του επιτρέψουν να καταστούν γνωστές στα κράτη-μέλη, να καταστούν γνωστέ από τα ίδια τα θέματα για να εξυπηρετηθεί ο τελικός στόχος, δηλαδή να διευκολυνθεί η πορεία του θύματος προς τις οργανώσεις αυτές που προσφέρουν βοήθεια. Και θα ήθελα επίση να αναφερθώ στην ε, ρήτρα για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Βρίσκεται στην ε, φάση της ε, υπογραφής και κύρωσης και τι σκοπεύετε να κάνετε ως προς την κύρωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Μπράντα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ορίζω και την Επίτροπο. Κάποιε ερωτήσεις έχω να κάνω για θέματα τα οποία θίξατε και εσεί οι ίδια. Καταρχάς, ό,τι αφορά την ίση αμοιβή. Είπατε ότι η έκθεσή μας κινείται προ τη σωστή ε, κατεύθυνση. Εμείς βασικά και προ εσά. Ε, ε, κινούμαστε. Ελπίζω να είναι η σωστή κατεύθυνση αυτή. Αναφερθήκατε και σε θέματα διαφάνειας που αποτελούν ε, το κλειδί της έκθεσής μας. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε καλύτερο νομοθετικό πλαίσιο προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν αναφερθήκατε σε μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, η περίπτωση της Ελβετίας, που έχει πραγματικά υποδειγματικό μοντέλο διαφάνειας και ίσης αμοιβή, ακόμα και για άτομα με, που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, όχι μόνο μεταξύ ανδρών και γυναικών δηλαδή. Έχουμε τα στοιχεία. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε άλλες μελέτες, άλλες έρευνες, προκειμένου να φτάσουμε στο επίπεδο που προβλέπουν οι συνθήκες της Ρώμης το 57. Και πέρα από τη διαφάνεια, πολλά στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκθεση και πιστεύω ότι πολλές γυναίκες περιμένουν από εσά να δείξετε το θάρρος, την τόλμη που χρειάζεται. Δεν ε, μπορείτε φυσικά εσείς να επηρεάσετε πολλά ε, όλες τις πτυχές της ίσης αμοιβή. Το ξέρουμε αυτό στη Γερμανία, για παράδειγμα, που υπάρχουν ε, οι, εθνικές, οι εθνικοί περιορισμοί, αλλά υπάρχουν τμήματα τα οποία μπορείτε να τα επηρεάσετε. Σας παρακαλώ λοιπόν να το πράξετε αυτό. Νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά τρομερό αν η απάντησή σας ήταν ότι δεν σκοπεύω να προωθήσω νομικές αλλαγές. Δεύτερο σημείο για την επόμενη Επιτροπή και σε ό,τι αφορά την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών ε, στην Επιτροπή Είχαμε την έκθεση σχετικά είναι, όπω ξέρετε ήταν πάρα πολύ καλή. Τι θα κάνετε λοιπόν για την ίση εκπροσώπηση στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα τελευταίο, τελευταίο σημείο για τι εξιστικέ διαφημίσει που θεωρώ ότι είναι σε άνθηση σε όλε τι χώρε. Ήταν πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο. Επί σειρά ετών ήταν αρκετά ποτική αυτή η τάση και τώρα έχει αλλάξει αυτό. σω θα έπρεπε να εξετάσουμε εκ νέου την νομοθεσία μα σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κουτάκη. ευχαριστώ την Επίτροπο που ήρθε. Όλοι εκτιμούμε τις επισκέψεις σα εδώ και το έργο σας για την Επιτροπή, τη δική μας. Είπατε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την ατζέντα μας και με άλλους επιτρόπους. Είναι πραγματικά εξαιρετική ιδέα. Ίσως θα έπρεπε ε, να καλούμε τακτικά και άλλους επιτρόπους και να τους ρωτάμε τι κάνουν και αυτοί Χαιρόμαστε ε, για το EPO ε, πώς ε, προωθήθηκε το θέμα αυτό και χαίρομαι που προχωράτε έτσι με το αστικό τμήμα και ούτω καθεξής. Πολλά πρέπει να κάνει η Επιτροπή μας, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι, ότι θα πρέπει να σεβόμαστε πάντα τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και σε κάποιες περιπτώσεις κολλάμε γιατί επισερχόμαστε σε τομείς που δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Θα πρέπει να δώσουμε τη φωνή που χρειάζονται οι γυναίκες σε θέματα FGM, εξαναγκασμένων γάμων, βίας κατά των γυναικών. Εκεί όπου μπορούμε να κάνουμε διαφορά. Συζητήσαμε ε, το θέμα ε, των ομοφυλόφιλων γυναικών στην, ε, στο Καμερούν και στην Αφρική. Για τις ποσοστώσεις τώρα. Πιστεύω ότι η συνάδελφος έκανε ένα μικρό λάθος, γιατί δεν είναι στην κυβέρνηση. Ο Κάμερον υποστηρίζει τις ποσοστώσεις, τις εξετάζει προσωρινές, προσωρινές ποσοστώσεις. Θεωρώ όμως ότι το θέμα των ποσοστώσεων είναι θέμα κρατών μελών που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά περίπτωση. Θα ήθελα να τονιστεί πιο πολύ η ε, εκπαίδευση Αναφερθήκατε στην αδιαμητρότητα. Ναι, κάτι θα πρέπει να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τρία στοιχεία τώρα. Θα πρέπει να είναι ευέλικτη, μη υποχρεωτική και βάση κρατούς μέλους. Μήπως όμως θα ήταν καλή ιδέα να συνέλθει μια ομάδα εργασίας από όλες τις ομάδες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Οκτώ άτομα δηλαδή λίγο πολύ, για να συζητήσουμε ποια είναι τα καθότητα ζητήματα για το Συμβούλιο και πού μπορούμε να κάνουμε μια υποχώρηση, γιατί νομίζω ότι στην παρούσα φάση θα πρέπει να κάτσουμε και να κοιτάξουμε τι ε, μπορούμε να θυσιάσουμε, γιατί πολλά θετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην οδηγία που θα τα χάσουμε και τα αγνοούμενα παιδιά. Ναι, 100% ε, σας υποστηρίζω. Ε, κάνω πάρα πολύ μεγάλο έργο προς την κατεύθυνση αυτή και προφανώς το Λίμανο Βασίλη έχει πάρα πολλά να πει. Ευχαριστώ. Λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λιωτάρτ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ σήμερα, να σας ευχαριστήσω και για την εισαγωγική παρατήρησή σας. Θα ήθελα πω ότι το 2011 ήταν το έτος για την ε, ενεργή γύρανση και για την ε, αλληλεγγύη μεταξύ των γενναίων. Ελπίζω να το γνωρίζετε αυτό. Ε, θα σας ενημέρωσα τώρα μόλις. Στην αγορά εργασίας υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες, πολλές ηλικιωμένες γυναίκες οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε πιο δυσχερή θέση. Το αναφέρατε. Ε, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών και το γεγονός ότι πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν διακριτική μεταχείριση στην εργασιακό τους βίο. Και συχνά, επειδή ε, είχαν ε, κάποιο κενό στο συνταξιδοτικό τους πρόγραμμα, αντιμετωπίζουν και προβλήματα φτώχεια σε προχωρημένη ηλικία. Υπάρχουν ε, λοιπόν πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα στο πρώτο πυλώνα και στις συντάξεις του πρώτου πυλώνα, στις ασφαλείς συντάξεις. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει σαφέστατη ε, διάκριση ε, σε ό,τι αφορά την ηλικία, αλλά και τη σύνταξη. Γιατί πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει νομοθεσία σε ό,τι αφορά ε, την διακριτική μεταχείριση βασιλικίας. Πώ μπορούμε λοιπόν να επιστήσουμε την προσοχή των γυναικών στο γεγονό αυτό και τι σκοπεύετε να πράξετε προ την κατεύθυνση αυτή επιπλέον. Προστίθεται το γεγονό ότι ε, πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν στερεότυπα σε ό,τι αφορά τα φύλλα. Πριν ε, από κάποιο καιρό η Εύα Μπριτ ε, Σβένσον κατέκτησε μια σχετική έκθεση. Θα ήθελα να ακούσω τι έχει γίνει με την έκθεση αυτή στι διάφορε γενικέ διευθύνσει. Έχω αποστείλει γραπτό ερωτήματα σε όλες τις γενικές διευθύνσεις ήταν πραγματικά λιπρό το αποτέλεσμα. Τι μπορείτε λοιπόν και τι προτίθεστε να κάνετε τον επόμενο καιρό προκειμένου σε όλους τους εργασιακούς τομείς να προτείνετε λύσεις για την καταπολέμηση αυτών των στερεοτύπων των φύλων, αλλά και για την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης των ηλικιωμένων γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκουμάη και κατόπιν στην κυρία Μπόσκουρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Πίτροπο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε εδώ. Θέλω να επικεντρωθώ σε κάποια σημεία, καθώς οι συνάδελφοι έθιξαν τα πολύ σημαντικά και θα ήθελα να ξέρω πότε θα έχουμε το σχέδιο προγράμματος του 2013, γιατί είναι καλό να έχουμε και διαφάνεια. Τώρα, για το ποσοστό της συμμετοχής των γυναικών στα συμβουλία. Νομίζω ότι σωστά τοποθετηθήκατε γι' αυτό σε ό,τι αφορά τη δεσμευτική νομοθεσία και τον κανονισμό θα πρέπει να ξεπεράσουμε τους χρονικούς και τους ποσοτικούς στόχους και να έχουμε αποτελεσματικές κυρώσεις αν δεν υπάρχει συμμόρφωση. Μιλήσατε για κατάλληλα μέτρα, πώς δηλαδή αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή και είμαι πάρα πολύ περήφανη γιατί όλοι οι φίλοι μου γνωρίζουν ότι από την παιδική μου ηλικία αγωνίζομαι για αυτό το θέμα και μου έχετε πολύ καλό εταίρο την κυρία Ρέντινγκ και δώστε τη μάχη αυτή γιατί είναι πάρα πολύ καλό για την οικονομία, για την κοινωνία και για όλους μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της ανεργίας στους νέους. Έχουμε φέτος ε, μία εκστρατεία Δημοκρατία ως Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και έχουμε μία εκστρατεία το μέλλον σου είναι το μέλλον και, το, και μιλάμε για μία εγγύηση για την ελληνική και βασίζεται σε ένα δημοκρατικό μοντέλο, είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τους νέους ότι όλοι και αναφερόμαστε στο ότι όλοι οι νέοι πρέπει να έχουν μία δουλειά και πρέπει να έχουν μία κατάρτιση. Κάναμε έναν υπολογισμό, είδαμε ότι χάνονται εκατοντάδες εκατομμύρια, αν έχουμε μία επένδυση 10 δισεκατομμυρίων, ε, τότε θα έχουμε 2,5 εκατομμύρια νέους με θέσεις εργασίας και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε και το θέμα αυτό και κατόπιν ε, σε ό,τι αφορά την εμπορία ανθρώπων ε, είχαμε μία σειρά προτάσεων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση στις περιπτώσεις που έχουμε και μεγάλες εκκλητικές εκδηλώσεις και ξέρω ότι και η Επίτροπος Μάλστρομ μαζί και με την Euro Europol, Eurojust και άλλους οργανισμούς που προσπαθούν να συντάξουν μία, ένα ε, πλήρες κείμενο για την καταπολέμηση της εμπορίας ε, και ε, κατά τη διάρκεια του Eurocup, του Ευρωπαϊκού Κυπέλου και για τους Ολυμπιακούς τι θα κάνει η Κομισιόν για να καταπολεμήσει το θέμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Εγώ πιστεύω ότι έχετε κάνει μία φανταστική εκστρατεία. Διασφαλίσουμε λοιπόν ότι είμαστε αρκετά ε, κάθετοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και χαίρομαι πάρα πολύ ε, που σας βλέπω εδώ. Είναι πάρα πολύ καλή στιγμή για λεγθέσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Μπόσκουρτ και κατόπιν κυρία Γιάροκα. you, uh, um, Ευχαριστώ. Τρία σχόλια. Καταρχήν ε, για τη δεσμή μέτρων για τα θύματα. Το Κοινοβούλιο θέλει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα φύλου και ε, χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για σας αυτό το θέμα. Σε ποιο βαθμό θα υποστηρίξει η Κομισιόν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως ε, σε ό,τι φορά τα μέτρα πρόληψης ε, και του εντοπισμού των συγκεκριμένων αναγκών, των θυμάτων και, και των αναγκών κατάρτισης για τους επαγγελματίες. Δεύτερον, θέλω να αναφερθώ στο θέμα της δεκτομής. Έχουμε μία μελέτη, όπως είπατε, βέβαια το 2013. Η Κομισιόν ε, θα παρουσιάσει μέτρα. Πότε θα πρέπει να αναμένουμε να παρουσίασε αποτελέσματα η Κομισιόν ε, για να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για το θέμα αυτό. Θα είναι το 2013 και η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με, για τη νέα σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Έχει ανοίξει τώρα στη στιγμή για τις υπογραφές. Ποια είναι τα σχέδια της Κομισιόν για την υπογραφή και, τη σύμβαση, και την κύρωση της σύμβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μας δώσετε τις νομικές αναλύσεις ε, σε μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Και ένα χρυσό αστέρι στην κυρία Πόσκα που σεβάστηκε ε, το χρόνο. Θα το σημειώσω στο ημερολογιό μου. Θα βάλω ένα χρυσό αστέρι δικά για σας. Λοιπόν, η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Γιάροκα και μετά η κυρία Τσέσκοβα. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε για τη δέσμευσή σας ε, να διατηρήσετε και τα θέματα της καταπολέμησης της ανέχειας ε, στην ημερησία διάταξη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ ε, που επεκτείνεται η στρατηγική για τους Ρωμά και σε άλλους Αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα θέλαμε να ε, μπορεί οπουδήποτε η Επιτροπή να έχει λόγο για τη συμμετοχή του Ρωμά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στα ευρωπαϊκά θέματα. Ε, έχουμε ένα σχέδιο δράση για του Ρωμά σε όλη την Ευρώπη. Σε ποιο βαθμό βλέπετε εμεί τα ευρωπαϊκά πολιτικέ ε, καταστάσει Ε, δημιουργούν ε, περικοπές ε, και σε προγράμματα για την καταπολέμηση της ανέχειας στις διάφορες χώρες. Σε ποιο βαθμό βλέπετε ότι το επιχείρημα της συμμετοχής του Ρωμά σε αυτές τις στιγμές της οικονομικής κρίσης που θίγει αυτά τα 40 εκατομμύρια άτομα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή και επίσης ε, τι θα κάνετε με την ε, εφαρμογή της οδηγίας και επίση είναι σημαντική αυτή η χρονική στιγμή για να δούμε ποιο πλήττεται από την κρίση και με ποιο τρόπο να ενδυναμώσουμε το σύστημα ε, κλιματική παρακολούθηση ε, και Επίσης, ε, να υπάρχει και συνεχής πολιτική δέσμευση. Αυτό που κατακτώσαμε να πετύχουμε τα τελευταία έτη, συνεχής πολιτική δέσμευση από τα τρία όργανα. Αυτή η πολιτική δέσμευση πρέπει να ενδυναμωθεί για να διασφαλίσουμε ότι και τα υπόλοιπα θέματα στα οποία αναφέρατε θα ολοκληρωθούν με επιτυχία. Όταν μιλάτε για την ερμοδιότητα λήψης αποφάσεων, Πρέπει να πιστήσω την προσοχή σα ότι όλα τα προγράμματα μείωσης της στόχιας ε, θα καταστούν ε, δυνατά και υλοποιήσιμα αν υπάρχουν καλοί ε, και αν υπάρχουν και άτομα νεότερες ηλικία αλλά και γυναίκες που να συμμετέχουν και να μπορούν να συμμετέχουν έτσι ώστε να κινηθούν και μικρότερες κοινότητες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό στο μοντέλο να δώσουμε και δύναμη ισχύει σε όσους ε, δεν μπορούν να μιλήσουν αυτή τη στιγμή και υποεκπροσωπούνται ε, σε καθημερινό επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Τσέσκοβα στη συνέχεια και μετά η κυρία Κοχμάιρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μα δίνετε να κάνουμε τη συζήτηση αυτή μαζί σα. Θα αναφερθώ αποκλειστικά στο θέμα των ποσοστώσεων και σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και σε άλλα τέτοια συμβούλια. Θα ήθελα να σα πω ότι στη τσεχική δημοκρατία από όπου και προέρχομαι ε, προωθείται και γίνεται αυτή η δημόσια συζήτηση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρώ ότι δεν θα μπορούμε να τις επιβαρύνουμε με ανελαστικές, ε, ανελαστικούς όρους για την ποσόστοση των γυναικών. Αυτό μπορεί να θίξει και ενδεχομένω μια γυναίκα, όπως ε, και έναν άντρα θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει περιττό γραφειοκρατικό άχθος σε ό,τι αφορά τις ε, υπόλοιπες μεγάλες ε, επιχειρήσεις. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα θέμα το πιο ποια εταιρεία θεωρείται μεγάλη ή μικρή στις διάφορες ε, χώρες. Αν επιμείνουμε στις ποσοστώσεις επισήμως και αν θεωρούμε ότι έτσι μπορούμε να αναγκάσουμε τις επιχειρήσεις, ε, μπορεί τελικά να ε, προωθήσουμε γυναίκες που δεν έχουν ουσιαστικέ αρμοδιότητες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί ε, προασπίζεστε τα δικαιώματα και ανδρών και γυναίκων. Θα ήθελα λοιπόν στο νομοθετικό σας έργο να δοθεί έμφαση σε όλες ε, τις πτυχές που θα μπορούσαν να συμφιλιώσουν ε, την οικογενειακή ζωή με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και κλείνω προκειμένου να μπορούν να αναλαμβάνουν επαγγελματικά καθήκοντα οι γυναίκες χωρίς να χρειάζεται να διακόπτουν την καριέρα τους. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που λαμβάνετε υπόψη τα σχόλιά μας. ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει Η κυρία Κοχμέριν και αν θέλετε λίγο πιο σιγά να μιλάτε για να μπορούν να σας παρακολουθούν και διερμηνείς. Ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, αλλά ήθελα να κάνω αυτή την παρατηρήση παρόλα αυτά. Thank you very much. Start. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρέντιν για την παρουσίασή σας. Ξέρετε ότι υποστηρίζω τα μέλα τα έτοιμά σας για ποσοστώσεις ε, στα δικαιωτικά συμβούλια, κυρίως ε, στη χώρα μου στη Γερμανία. Είναι ένα ιδιαίτερα επίμαχο ζήτημα, αλλά σας ε, παρακαλώ να είστε κάθετοι σε αυτό και θέλω να τονίσω κάτι ακόμα σήμερα. Στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών ε, εγκρίναμε ε, την γνωμοδότησή μας για τον κανονισμό για το προσωπικό και επικεντρωνόμαστε σε θέματα γυναικών φυσικά εδώ και Φυσικά βλέπουμε ότι όσο ψηλότερα ανεβαίνουμε στην ιεραρχία, τόσο λιγότερε είναι οι γυναίκε και θέλουμε να αλλάξει αυτό. Και υπάρχουν και πάρα πολλά μέτρα για τι συμφιλίε τη επαγγελματική και τη οικογενειακή ζωή, αλλά κυρίω ε, αυτά ε, έχουν να κάνουν με τι γυναίκε. Ε, γονική άδεια 80% τη λαμβάνουν οι γυναίκε και αυτό σημαίνει ότι διακόπτεται στη διδρομία των γυναικών. Και γιατί οι άνδρε δεν παίρνουν γονική άδεια, θέλουμε να αλλάξει αυτό και θέλουμε και εκεί να έχουμε ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Εμείς ε, γνωρίζουμε ποιες ε, είναι, ε, ποια είναι τα όρια του προϋπολογισμού, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν την πολιτική αξιοπιστία. Αν ζητάμε από τα κράτη-μέλη να εισαγαγούν συστήματα για τη γονική άδεια και εμείς πρέπει να το κάνουμε. δηλαδή αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε πώς οργανώνεται η γονική άδεια ε, του, η άδεια πατρότητας ε, και ε, σήμερα βλέπουμε μια σημαντική μείωση ε, στο εξάμεινο και θέλουμε να έχουμε 60 της 100 του προηγούμενου μισθού μέχρι ένα ανώτατο ποσό που να είναι πιο κοντά στο πραγματικό κόστος που έχει ένας νέος γονιός. Και φυσικά θα πρέπει να περάσει αυτό το θέμα και από άλλε επιτροπές, θα περάσει και από την Ολομέλεια. Αλλά θέλουμε να ζητήσουμε την υποστήριξή σας από αυτού και, να ελπίζουμε ότι η Κομισιόν θα ευνοήσει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και... Έχουμε ακόμα ένα συνάδελφο, μία συνάδελφο, την κυρία Σαββόρσκα που θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρατηρήσεις. Μέχρι στιγμής πιστεύω δεν απάντησε κανείς στη δική σας ερώτηση. Πώς δηλαδή διαβλέπουμε τη συνέχεια για την οδηγία για τη μητρότητα. Η κατάσταση όπως τη βλέπω εγώ σε ορισμένα κράτη-μέλη όπου η προστασία των γυναικών ως ε, εγγύων ή λεχουσών γυναικών ε, από το χώρο εργασίας ε, δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Πρέπει να δούμε λοιπόν ε, την κατάσταση. Η κυρία Στρελαστικός δεν είναι εδώ, αλλά θα πρέπει ίσως να κοιτάξουμε εάν διαδικαστικά είναι προτιμότερο να καταρτιστεί ρέον κείμενο της οδηγίας όπου θα γίνεται λόγο και για πατρική άδεια, αλλά από ταυτόχρονα θα πρέπει να αλλάξει και ο τίτλο τη οδηγία. γιατί εφόσον μιλήσουμε για άδεια για τον πατέρα, δεν μπορούμε μόνο να μιλούμε για προστασία της εγκύου στον χώρο εργασίας. Δεν βλέπω τι άλλη λύση θα μπορούσαμε να έχουμε για να διαφύγουμε από την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν, δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα αυτό. Η κυρία Στρέλα όμω δεν είναι σήμερα εδώ. Πάντω η επίτροπο. θα πρέπει να γνωρίζει ότι είμαστε ήδη στο τέλος μιας σειράς ε, συνομιλιών με την Προεδρία της Δανίας με την υποστήριξη και της κυρίας Εστρέλα και των συντονιστών μόνο να πέστειλε η κυρία Εστρέλα μια επιστολή Προ το Συμβούλιο λέγοντα ότι είμαστε διατεθειμένοι να συστήσουμε τα εκκρεμή ζητήματα. Προσπαθούμε δηλαδή να επισημάνουμε ότι εμεί το ρόλο μα τον βλέπουμε επικοδομητικά. Θέλουμε να έχουμε επικοδομητικό ρόλο, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει όμω από την Προεδρία λάβαμε μια απάντηση που έλεγε ότι πολύ ευχαριστώ να συστήσουμε τα θέματα αυτά. Μέχρι εκεί όμως πρέπει να περιμένουμε δηλαδή να δούμε ποια συγκεκριμένη εξέλιξη θα έχει η υπόθεση αυτή. Θα προσπαθήσουμε πλευρά μας να επιλύσουμε αυτήν την ε, ε, κατάσταση. Το λόγο εσείς παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επανέλθω μέσω στο θέμα της ε, άδειας μητρότητας πατρότητας και να απαντήσω ότι είναι πολύ δύσκολο βέβαια να περάσουμε στο θέμα της άδεια πατρότητας εφόσον δεν έχει επιληθεί ακόμη άδεια Με χαρά ακούω ότι το Κοινοβούλιο έχει εκδηλώσει ευελιξία, ότι η Προεδρία της Δανίας από πλευρά τη, ε, δήλωσε πως θα εκθέσει το ζήτημα στο Συμβούλιο στους υπουργού, βεβαίω και εγώ θα προσπαθήσω και πάλι να συνομιλήσω με την Προεδρία της Δανίας και κάθε φορά που βλέπω υπουργό, κάθε φορά που επισκέπτομαι κράτος μέλος, ε, θέτω το ζήτημα και πάλι. Αλλά σας ε, διαβεβαιώ ότι δυστυχώς δεν έχουν ε, πολύ όρεξη του Συμβούλιο να το συστήσουν το θέμα αυτό ανοιχτά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ και ελπίζω πάντα ότι και οι δύο πλευρές θα επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την ελπίδα ότι η διαπραγματεύσεις σημαίνουν και υποχώρηση ως προς κάποιες θέσεις για να εξασφαλίσουμε κάποια πρόοδο. Και τότε και η πρόταση της κυρίας Αμπόρσκα ασφαλώς θα τεθεί επί της τράπεζας των διαπραγματεύσεων. Αλλά όσο δεν υπάρχει τράπεζα διαπραγματεύσεων και όσο κάθεται κανείς γύρω από αυτήν την τράπεζα δεν, έχει, ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Για τα προγράμματα. Στα νέα προγράμματα το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2013-2020, όπως γνωρίζετε, περιλαμβάνει τα συγχωνευμένα, συγχωνευμένα έξι ε, προγράμματα που έχουν συγχωνευτεί σε δύο. Έχουμε το πρόγραμμα για την Ιθαγένεια, το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα δύο προγράμματα. Χάνονται τα ονόματα λοιπόν, οι τίτλοι, αλλά δεν χάνονται οι, δεν οι στόχοι και οι στόχευση των προγραμμάτων αυτών. Ε, τα κονδύλια παραμένουν λίγο πολύ τα ίδια. Έχω καταφέρει δηλαδή να διαφυλάξω, να διατηρήσω το επίπεδο της χρηματοδότησης. Καθώς είμαι λοιπόν επίτροπος αρμόδια για την ε, δικαιοσύνη, μπορώ τα κονδύλια από το πακέτο της δικαιοσύνης να τα διαθέσω στην προστασία των γυναικών σε τέτοιες περιπτώσεις όπου έχει ασκηθεί βία κτλ. Δηλαδή έχω μια ευελιξία ως προς το θέμα αυτό, δηλαδή από τη δικαιοσύνη μπορώ να προστατέψω, χάρη στη δικαιοσύνη μπορώ να προστατέψω τα δικαιώματα των θυμάτων. Τα θύματα δε το είναι γυναίκες, θύματα βίας και έτσι μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Διαφορετικοί λοιπόν τίτλοι, αλλά συγχωνευμένες δράσεις και πιο απλουστευμένη χρηματοδότηση για τον δικαιούχο. Περισσότερη συνεργατική δράση, εστίαση καλύτερη και έτσι και για την κυρία Γιαρόκα, μπορούμε να ε, ενσωματώσουμε και ανάγκες συγκεκριμένη πολιτικής που μπορούμε να αναπροσδιορίζουμε σύν το χρόνο. Είδατε παραδείγματι τι καταφέραμε με τους Ρωμά. Αντιμετωπίσαμε, προσκρούσαμε πάνω στο πρόβλημα των Ρωμά Προσπαθούσαμε να βρούμε ψίχουλα για να βοηθήσουμε και να προχωρήσουμε προς μία λύση. Και τώρα με το νέο πρόγραμμα Ίσης Ευελιξία μπορούμε, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, εφόσον θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, να αναλάβουμε τη σχετική δράση. Πάντως ε, το ζήτημα και η δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ως προς τη χρηματοδότηση των πρωτοβουλειών για τους Ρωμά ήταν ένα πολύ καλό δίδαγμα. Είδαμε ότι ήταν πολύ α, ανελαστικές οι διατάξεις. Μην ανησυχείτε λοιπόν, υπάρχουν ήδη κάποιες δυνατότητες, έχουμε υπόψη μας διασυνοριακές δράσεις, ο προϋπολογισμός διατηρείται λίγο πολύ και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Για το FGM, μαζί με το Ινστιτούτο αναπτύσσουμε αυτή τη χαρτογράφηση ε, του θέματος της κλειτοριδεκτομής ε, με ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δρούν και έξω από την Ευρώπη, ε, ε, ο Επίτροπος Αρμόδιος για την Αναπτυξιακή Βοήθεια και την Κατεπίγουσα Βοήθεια έχουν ε, την υπόθεση αυτή στην κύρια πρώτη, στις κύριες προτεραιότητες τους, αλλά το θέμα που έχουμε εμείς να επιλύσουμε είναι ένα εσωτερικό ευρωπαϊκό πρόβλημα και άρα είναι πολύ σημαντικό το Ινστιτούτο να μας δώσει αυτήν την χαρτογράφηση, αυτή την καταγραφή της κατάστασης για να δούμε πού παρουσιάζονται μεγαλύτερα οξυμένο χαρακτήρα τα προβλήματα. Εγώ έκθεση από το Ηνωμένο Βασίλειο ή που να αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχω δει μάλλον ούτε και εσείς. Παρακαλώ ενημερώστε μας, δώστε μας ό,τι στοιχεία έχετε για αυτή την έκθεση για να την μελετήσουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δύο φορές την ίδια δουλειά. Εάν έχετε κάποια στοιχεία θα προσπαθήσουμε να τα ενσωματώσουμε. Αν έχει ήδη γίνει κάποια μελέτη δηλαδή. Εν γέννη, για το θέμα της βίας, τα δύο Ινστιτούτα συνεργάζονται και ήδη έχω ζητήσει από την αρχή, από τη Βιέννη, να προσφέρει χείρα βοηθείας στο Βίλνιους για να προχωρήσει και το Βίλνιους. Και το Βίλνιους προχωράει καλά βέβαια. Έχει περίπου 40 μέλη ε, προσωπικού, 40 υπαλλήλους ε, αναπτύσσει ενδιαφέροντα ευρήματα στο ζήτημα της ισότητας των φύλων ήδη και μπορούμε να πούμε ότι θα έχει μπει σε, ε, στην τακτική του ε, δουλειά, στην ταχύτητα κουραζιέρα, όπω λέμε το 2013. Θέλουμε λοιπόν να συνεργάζονται τα Ινστιτούτα, αλλά όχι να επικαλύπτει το ένα τη δουλειά του άλλου. Έχουν διαφορετικέ δυνατότητε και αν συνεργαστούν καλά μπορούν να έχουν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά ε, τη δυνατότητα να επιτελέσουν τη δουλειά του. Ένα παράδειγμα, το Ινστιτούτο για τα φύλλα, για την ισότητα των φύλων, όχι απλώ ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι ένα Ινστιτούτο το οποίο ανήκει στην Επιτροπή και στην Επιτροπή σα, στην Κοινοβουλευτική σα Επιτροπή. Είναι ένα Ινστιτούτο το οποίο ε, κάνει δουλειά που απευθύνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά όλε τι πολιτικέ που χαράζονται. Δηλαδή δεν ε, ασχολείται μόνο με τη διάσταση των φύλων. Ε, επί παραδείγματι τώρα έκαναν μια δουλειά, μια μελέτη για τις κλιματικές αλλαγές και την επίδρασή τους στην ε, γυναίκα, στις γυναίκες. Επίσης είχα την ευκαιρία και σε ένα πρόγευμα με τον πρόεδρο να συζητήσω το θέμα αυτό, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει όχι μόνο ε, η μία επίτροπος, αλλά όλοι οι επιτροποί, γιατί όλοι οι επιτροποί έχουν υπογράψει το χάρτη και άρα είναι όλοι συνυπεύθυνοι και τα θέματα τα οποία εσείς ανακοινήσατε εδώ ως προς τα χαρτοφυλάκια διαφορών επιτρόπων, φερειπίν φτώχεια, νεολαία, ανεργία, όλα αυτά τα ζητήματα. Προφανώς και μάλιστα κύριε Πρόεδρε παρακαλώ προσκαλέστε κι εσείς, όποτε θεωρείτε σκόπιμο, άλλους επιτρόπους να σας συζητήσουν στο πλαίσιο των δικών τους χαροφυλακίων θέματα ισότητας των φύλων. Και χάρη στην ευκαιρία αυτή πιστεύω θα μπορέσετε και να τους ευαισθητοποιήσετε περισσότερο στις ανάγκες των γυναικών και των γυναικών βέβαια σε θέσεις ε, προβεβλημένες. Αυτά λοιπόν ε, οι διαβουλεύσεις θα συνεχίσουν έως τα τέλη Μαΐου. Από ό,τι βλέπω γιατί έχουμε λάβει τεράστιο όγκο προτάσεων με πολύ ε, συγκρόμενες μερικές φορές θέσεις. Πολλά θέματα θα προκύψουν ως προς το περιεχόμενο και έτσι όταν ολοκληρωθεί αυτή η συλλογή του υλικού έως το τέλη Μαΐου θα γίνει η ανάλυση πολύ προσεκτικά και θα προτείνουμε μία δράση προς τους επιτρόπους που θα ήθελα να μεταφραστεί σε ένα νομοθέτημα. Και στο οποίο θα χρειαστώ τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να μιλάω σαν το Σαρκοζή τώρα, δεν είμαι σε τέτοια απόγνωση, αλλά πραγματικά χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Γιατί πρέπει σε κάθε επίτροπο που συναντάτε να μιλάτε, να τον σταματάτε στον δρόμο και να του λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κοινοβούλιο. Εγώ ξέρω πόσο σημαντικό είναι το θέμα για το Κοινοβούλιο, αλλά εάν συναντήσετε κάπου κάποιον επίτροπο, μη λησμονήσετε να τον αναφέρετε. Γιατί θα έχουμε μετά και τη διελκυστήνητα για τις ποσοστώσεις στο επόμενο στάδιο. Επίσης, για τον κανονισμό ε, υπηρεσιακής κατάστασης τώρα. Ε, μπορώ να πω μόνο ότι έχουμε θίξει και έχουμε θέσει σε υψηλό επίπεδο προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων, την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων. Ε, υπάρχουν στόχοι, οι συζητήσεις για ποσοστώσεις, σχεδόν φτάνουμε στους στόχους που είχαμε ορίσει για, το, για τα μέσα μεσαία στελέχη έχουμε 30% στόχο για την Επιτροπή δεν έχω μαζί μου στοιχεία ακριβή, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο 37-38%. Έχουμε επομένως 27-28%. Ε, Άρα πλησιάζουμε το 30% τον στόχο μας ε, σε πολύ λίγο καιρό και υπάρχει και το σχετικό φυλάδι για όποιον ενδιαφέρεται να μελετήσει την κατάσταση και την πρόοδο. Στόχος είναι και να προάγονται όσο δυνατόν περισσότερες γυναίκες στην ανώτερη διοίκηση η γενική μου διεύθυνση δυστυχώς δίνει πολύ κακή εικόνα γιατί υφίστανται διακρίσεις οι άνδρες Εν πάση περιπτώσει όμω, ε, πρέπει <laughs> να ομολογήσουμε ότι με τον πρόεδρό σα έχουμε κάποια εξισορρόπηση των φύλων. Έχω 60% των γυναικών ε, στη, στα μεσαία στελέχη και στα ανώτερα 80% γυναίκε. Άρα μάλλον αδικούμε τους άντρες. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό όμω δεν είναι αστείο, είναι πραγματικότητα. Για, και αυτό σα δείχνει πιστεύω ότι όταν κανείς αναζητεί γυναίκε με ταλέντο, με ικανότητε, τι βρίσκει, υπάρχουν. Άρα το ζήτημα είναι αν κανείς πράγματι αναζητεί, εάν θέλει να βρει γυναίκες μετανάστες. Διότι αυτό που θέλουμε είναι να προαγάγουμε γυναίκες με δεξιότητες, ικανές, όχι απλώς να τοποθετούμε σε μια θέση μια γυναίκα μόνο και μόνο λόγω του φίλου της, γιατί εκεί θα τελειώσει και η ιστορία. Ε, πρέπει πάντοτε να αναζητούμε τις πιο ικανές γυναίκες, γυναίκες με τις πιο πολλές δεξιότητες και όχι βέβαια να ε, επιβάλλονται διακρίσει βάρο των ανδρών μόνο και μόνο γιατί έχουμε αποφασίσει να προαγάγουμε τι γυναίκε ή να προωθήσουμε τι γυναίκε. Για το ζήτημα των Ρωμά είναι ένα καθόδο ζήτημα, ένα δύσκολο ζήτημα όπω γνωρίζετε. Το γεγονό ότι οι πρωθυπουργοί υπέγραψαν δέσμευση ότι θα εισαγάγουν τις στρατηγικές για τους Ρωμά, μας βοηθεί να θέσουμε στην τράπεζα, να τοποθετήσουμε στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων προτάσει για του Ρωμά. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τώρα τη συζήτηση. Σε μερικέ εβδομάδε μόνο πιστεύουμε ότι θα έχουμε προτάσεις για εθνικέ στρατηγικές και αναλύσεις των προτάσεων αυτών και φυσικά παρακολουθούμε την κατάσταση εκ του σύνεγγυ και θα έχουμε και τη δυνατότητα εάν χρειαστεί τη χρηματοδότηση να την διαθέσουμε έτσι ώστε να ε, φτάσουμε στο σωστό στόχο. Αλλά υπάρχουν εθνικές στρατηγικές για τους Ρωμά. Δηλαδή το κύριο βάρος για την ανάληψη δράσης ε, στο θέμα της ε, κοινωνικής ενσωμάτωσης στα σχολεία κτλ. ανήκει στα κράτη-μέλη. Βία. Συνολικά. Ξέρετε, ότι δεν είμαι φίλος γραφειοκρατίας. Ξέρετε ότι ιδιαίτερος προτιμώ να έχω συγκεκριμένη δράση, συγκεκριμένα αποτελέσματα και πράξεις. Γι' αυτό έχω και την πρόταση μέτρων, το, τη δέσμη μέτρων για τα θύματα που έχει ουσία, που έχει ζουμί, γιατί μπορούμε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα μέτρα, όχι απλώς γενικόλογες ιδέες. Η προστασία των θυμάτων έχει ζουμί, σάρκα και οστά και άρα μπορούμε να δώσουμε ουσιαστική προστασία στα θύματα και λύσεις. Επίσης, τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης, το ευρωπαϊκό έτος του πολίτη, της ταγένειας, μπορούμε πιστεύω να το συνδυάσουμε με όλα αυτά που κάνουμε για τους πολίτες και με την ευαισθητοποίηση στο θέμα της βίας εις βάρος των γυναικών. Που αποτελεί μια κύρια και σοβαρή προτεραιότητα για τον τρόπο που εργαζόμαστε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Παρβάνοβα για τη δική της ε, στάση ε, στην υπόθεση αυτή. Θα ήθελα να πω ότι κάνουν ό,τι μπορούν οι ειδικοί μας για να ετοιμάσουν το καλύτερο δυνατό κείμενο, νομοθετικό κείμενο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι πρόκειται για μια πρώτη απόπειρε με αυτόν τον τρόπο για παραγωγή νομοθετήματο ευρωπαϊκού. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιτύχει και πιστεύουμε ότι θα επιτύχει και ότι θα έχει και πολλά αντίστοιχα ε, παραδείγματα στο μέλλον. Για την σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ε, καταπολέμηση της βίας βάρος των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας αναλύουμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά Ξέρετε, δεν είναι απλώς να πούμε υπογράφουμε μια σύμβαση. Αυτό είναι μια νομική πράξη. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν αυτό να το κάνουμε ε, χωρίς προσεκτική ανάλυση, χωρίς πραγματική μελέτη των συνεπειών αυτής της υπογραφής, άρα οι νομικές μας υπηρεσίες, οι νομικοί ειδικοί ε, τα, τι μελετούν. Θα ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη στο τέλος του έτους και θα σας ενημερώσω βεβαίως όταν θα έχω συγκεκριμένα στοιχεία για τις προτάσεις των πραγματογνωμόνων μας. Κάτι που λησμόνισε και φορά τους πολίτες. Ξέρω το 2013 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος του Πολίτη, των πολιτών. Δηλαδή, Δηλαδή θα έχει συγκεκριμένες δράσεις, ε, θα παρουσιάσει συγκεκριμένες δράσεις ε, και τα όσα πράττει για τον πολίτη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι τα οράματα του πολίτη, τι θέλει ο πολίτης να κάνουμε, πώ πώς θέλει να αλλάξουμε πολιτικές. Ο δημόσιος διάλογος λοιπόν που θα αναπτυχθεί θέλω να έχει διαφορετική φύση. Στις 9 Μαΐου δημόσιος διάλογος, διαβούλευση με τον πολίτη, ώστε ο πολίτης να μας πει τι θέλει να καλύψει το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών, τι θέλει να, τους να του προσφέρει, τι θέλει να περιλάβει το έτος των πολιτών ως θέματα. Γι' αυτό παρακαλώ και εσείς να είστε ενήμεροι και σε επαγρύπνηση. Στις 9 Μαΐου θα έχουμε αυτή την δημόσια διαβούλευση για το έτος των πολιτών. Μην ξεχνάμε ότι το 50% των πολιτών είναι γυναίκες και θέλουμε όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα να προετοιμαστούν οι πολίτε και να βοηθήσουν την προετοιμασία αυτού του Ευρωπαϊκού Έτου των Πολιτών και βεβαίω θα, θα ε, εκπονηθεί και η Ευρωπαϊκή η έκθεση για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Προσπαθούμε με διάφορα στοιχεία λοιπόν που θα προκύψουν από το έτος αυτό ε, να ε, καλύπτουν γυναικών κατά τρόπο αποτελεσματικό. Οι αποκλήσεις μισθολογικές ανάλογα με το φύλλο. Ξέρετε ότι αποτελούν ένα περίπλοκο ζήτημα. Έχουν πολύ περίπλοκες διαστάσεις και κυρίως για λόγους νομικούς. Γιατί ναι μεν υπάρχει, υπάρχουν οδηγίες οι οποίες απαγορεύουν ε, την ε, καταβολή διαφορετικών μισθών ε, για την ίδια εργασία και άρα κανείς μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια χάρη σε αυτές τις οδηγίες. Αλλά το ζήτημα που έχουμε κυρίως είναι ε, άλλες μορφές εργασίας όπως η ε, μερική απασχόληση και άλλες μορφές εργασίας και άρα θα πρέπει να συζητήσουμε και με τον Επίτροπο των Αρμόντων για τα κοινωνικά ζητήματα για να δούμε το κύριο και σοβαρότατο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε ως προς τη φτώχεια των γυναικών στην, ε, στα γυρατιά. Ε, που είναι άμεσα σχετιζόμενο και με τη μέρημνα, με τη φροντίδα για τα παιδιά και γενικότερα με την παροχή φροντίδας για όποιον έχει ανάγκη είτε είναι παιδιά είτε είναι ηλικιωμένοι. Οι γυναίκες θα βρεθούν ε, και σε ε, προχωρημένη ηλικία να έχουν κακή υγεία και να αντιμετωπίσουν το φάσμα της φτώχειας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και με τον Επίτροπο των Αρμόδιο για τα κοινωνικά θέματα να έχετε την ευκαιρία, να φροντίσετε να βρείτε μια ευκαιρία να συζητήσετε το θέμα αυτό συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη διαφάνεια, για το θέμα της διαφάνειας. Όπου επίσης βλέπουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και με τους ε, εργοδότες με το χώρο της παραγωγής, με τη Γερμανία, την Αυστρία, την, Πολο... την Πορτογαλία. Ε, ήδη έχουμε κάνει κάποια βήματα προόδου, καταγράφουμε ποια είναι η κατάσταση και κυρίως τι είδους αλλαγές σημειώνονται. Και ίσως με τους υπουργού από αυτές τις κυβερνήσεις, τους αρμόδιους για την διαφάνεια, για τους κανόνες περί μπορούμε να συζητήσουμε και να μάθουμε από αυτούς σε ποιον απευθύνονται όταν χρειάζονται κάποια στοιχεία. Απευθύνονται στην ηγεσία των μεγάλων επιχειρήσεων, μιλούν μόνο με μεγάλες επιχειρήσεις, μιλούν και με μικρομεσαίες. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το διαρευνήσουμε και μέσω των Υπουργών για να προχωρήσουμε στην υπόθεση αυτή για τη διαφάνεια. Κοιτάω πολύ γρήγορα, Πρόεδρε, αν έχει μείνει τίποτα που δεν απάντησα. Την είπα την κλειτοριδεκτομή, την κάλυψα νομίζω. Τι έμεινε. Ναι, θα σας ενημερώσω. Δεν ακούστηκε η κυρία Γκουρμάη. Δυστυχώς. Ε, θα σας ενημερώσει η ομάδα μου που επεξεργάζεται θέματα αυτά. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι κάλυψα τα κύρια ε, ερωτήματα. Αν τυχόν λησμόνησα κάλλη, ασφαλώς θα με θα μου το υπενθυμίσει η γραμματεία σας και θα σας απαντήσω γραπτός. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ την κυρία Ρέντινγκ. Όπως ε, γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία σας ε, στην Επιτροπή αυτή, το να έχουμε την δυνατότητα να μας παρουσιάσετε το πρόγραμμα που σχεδιάζει η Κομισιόν. Ε, έτσι λοιπόν, να κάνω και εγώ δύο σχόλια. Ξέρουμε ότι δίνεται μεγάλη σημασία στα θέματα αυτά και ενδιαφέρεστε πάρα πολύ να παρευρίσκεστε εδώ. Αλλά είπατε ότι θα συναντηθείτε και με άλλου επιτρόπου και εμεί θέλουμε να συναντηθούμε με άλλου επιτρόπου και είναι σημαντικό να δούμε τα θέματα αυτά μαζί του, γιατί τα θέματα αυτά αφορούν πολλού τομεί πολιτική και Προσπαθούμε να οργανώσουμε συναντήσεις και με άλλους επιτρόπους, αλλά όπως είπατε και εσείς είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό, γιατί τα θέματα της ισότητας των δύο φύλων είναι ουσιαστικά θέματα που άπτονται διάφορων ε, πολιτικών και επίσης συμφωνούμε σε ό,τι αφορά τους ε, δωρεούς οργανισμούς και τον οργανισμό στο Βιλνούς ε, και το ΕΦΕΓ είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη τα θέματα που αναφέρουν αυτοί οι οργανισμοί και να διασφαλίζουμε την βελτίστη δυνατή συνεργασία. Η συνεργασία λοιπόν είναι το σημείο κλειδί. Συμπερασματικά λοιπόν, θα έλεγα να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον επικοδομητικό διάλογο στο μέλλον. Όπως είδατε υπήρχαν ε, πάρα πολλές ερωτήσεις από τους βουλευτές, ε, ενδιαφέραν πάρα πολύ τους συναδέλφους, τα όσα είπατε και σας ευχαριστούμε και πάλι που παρευρεθήκατε εδώ. Okay, or... vill Bara fortsätta mötet och det är inte så mycket. Θα ήθελα να συνεχίσουμε με τη συνεδρίασή μας. Δεν έχουμε πάρα πολλά θέματα που να έχουν απομείνει στην ε, ημερήσια διάταξη. Το σημείο 20 το συζητήσαμε όταν ε, είχαμε χρόνο πριν την έλευση της κυρίας Ρέντινγκ. Μας έχει μείνει μόνο το σημείο 21, τα διάφορα και δεν υπάρχει κάτι από τα διάφορα. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο 22, το τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης και αφορά τις ημερομηνίες για την επόμενη συνεδρίαση. 29 και 30 Μαΐου ήταν ημερομηνίες που είχαμε σχεδιάσει, αλλά τώρα θα συναντηθούμε μόνο στις 30 Μαΐου. Αυτή είναι η τελευταία ημερομηνία που ορίσαμε, 30 Μαΐου μόνο. Θα συνεδριάσουμε και εδώ να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση και θέλω να σας ευχηθώ καλό απόγευμα.